Bene colleghi, possiamo... Non funziona? Sì, ma non, non, non, è, non, non, è non si sente. Colleghi, per favore, prendete... Sì, Συνάδελφοι, καθίστε. Όπως προβλέπετε, θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Καθίστε παρακαλώ, μην καθυστερούμε. Για την ψηφοφορία την σχετική με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Ετοιμάστε την ηλεκτρονική σας κάρτα παρακαλώ. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε αρκετές και περίπλοκες ψηφοφορίες μπροστά μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ καθίστε, μην αργείτε. γιατί μετά έχουμε επίσης και την υπόλοιπη μέρη διάταξη, η οποία είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη. Λοιπόν, καθίσατε όλοι όπως βλέπω. Η έκθεση του κυρίου Μποντής πρώτη. Θα ξεκινήσουμε με την παράγραφο 1 και την τροπολογία 21. και είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ Δεκτή. Συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κοντράρι. Andiamo all'emendamento 28. Περνάμε στην 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 36 πλέον. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 43 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 72 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή τοπολογία 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Περνάμε στη 12. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν καταλαβαίνω το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για τη 14. Ψηφίζεται ηλεκτρονικά την 14. Τρεις δεν ψήφισαν, εν πάση περιπτώσει τέλος της ψηφοφορίας 30 κατά 33 υπέρ. Η κυρία Λούνατσεκ. Ψηφίζω υπέρ, δεν λέει η κυρία Λούνατσεκ, δεν έχω κάρτα μαζί μου. Λοιπόν, δεκτή. Η 17. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 20. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή τώρα έχουμε τις νομοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας με την 2 ξεκινάμε ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή η 3 υπέρ κατά Αποχές δεκτή. Για μια στιγμή. Μπορούμε να ψηφίζουμε ομαδών σε εισαγωγικά από την 5 μέχρι και την 9. Διαφωνεί κάποιος? Όχι. Συνεπώς λοιπόν ψηφίζουμε 5 με 9 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Εφόσον συμφωνείτε θα κάνουμε το ίδιο πράγμα από την 11 μέχρι και τη 14. Λοιπόν, έχει κάποιο αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Περνάμε στην 16. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία τελική. Ξεκινάμε. Λοιπόν, 68 ψηφίζονται, 63 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές, συγχαρητήρια ε, στον εισηγητή. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος για την διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Μαυροβουνίου. Ο κ. Στάνοκ είναι ο εισηγητής. Ξεκινώ με την τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία προφορική 2 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τώρα η κανονική 2 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Η 3 υπέρ, κατά, αποχές δεκ, απερίφθη. Η 4 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 5 υπέρ. Α, εδώ έχει ζητηθεί ηλεκτρονικός έλεγχος για την 4, λέει ο πρόεδρος. Ψηφίζουμε λοιπόν την 4 ηλεκτρονικά. Λοιπόν, 67 ψηφίσαντες, 61 υπέρ, 6 κατά, 0 αποχές. Οι 5 λοιπόν τώρα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, μερσή. Η 6 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε στην 12 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 14 υπέρ, κατά, Αποχές δεν φαίνεται εύκολα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 14. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 14. 66 ψηφίσαντες. 48 όχι 17 ναι απορρίπτεται. Λοιπόν 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά δεν φαίνεται καθαρά το αποτέλεσμα ηλεκτρονική ψήφος για την 25 ξεκινάμε 67 ψηφίσαντες, κάποιοι δεν ψηφίζουν, 70 είναι οι κάρτες οι οποίες είναι στο μηχάνημα. 29 όχι, 38 ναι. Λοιπόν, 26 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 27 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 28 απεσύρθη, 29 με τροπολόγηση προφορική υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά δεν φαίνεται καθαρά το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε την 36 ηλεκτρονικά. Εβδομήντα κάρτες λοιπόν λέει ο πρόεδρος, 64 ψηφίσαντες. Κάποιοι συνάδελφοι είναι πολύ αφηρημένοι. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας 29 κατά 38 ναι. 37 τώρα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απερίφθη το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικός έλεγχος α όχι έλεγχος στο 41ο τμήμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία στην 41ο τμήμα. Ψηφίζεται. Κάποιοι συνάδελφοι παραμένουν αφηρημένοι. Λοιπόν, 38 υπέρ, 28 κατά, δεκτό το πρώτο τμήμα, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, Αποχές δεκτό. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην προφορική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική 4 υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο για την 4 την προφορική 4 διευκρινίζω 71 κάρτες, 63 ψηφίσαντες. 31 κατά, 30 υπέρ. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 69 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεύτερο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας 69. Ξεκινάμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, 69 ψηφίσαντες. 33 όχι, 36 ναι, δεκτή. Η συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 73 υπέρ, κατά, Λοιπόν, δεν είμαι βέβαιος. Ξεκινάμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 73, την προφορική τροπολογία. 70 κάρτες στο μηχάνημα, λέει ο πρόεδρος. Επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 73 με την προφορική τροπολόγηση. Πέρας της ψηφοφορίας. 32 κατά 34 υπέρ δεκτή. Το 74 τώρα. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 76 υπέρ. Κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 76. Ψηφίζουμε. Για την 76. Τέσσερις συνάδελφοι δεν δέχονται να ψηφίσουν. Λοιπόν, μειώνεται ο αριθμός τους βέβαια. Λοιπόν, 30 κατά 36 υπέρ δεκτή αιτιολογική σκέψη α, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονική ψήφος, τελική, άρχεται η ψηφοφορία. Για να δούμε, θα ψηφίσετε όλοι στην τελική ψήφο. Όχι, πάντα δύο συνάδελφοι δεν ψηφίζουν. Λοιπόν, 62 υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές συγχαρητήρια στον εισηγητή. Όλα πήγαν καλά μέχρι τώρα. Περνάμε τώρα στην πιο δύσκολη ψηφοφορία και περίπλοκη ψηφοφορία η έκθεση Oman Reuten. Θέλετε να λάβετε το λόγο προηγουμένω. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εφέτος είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει μια άποψη η οποία να είναι εξισορροπημένη. Γιατί όπως ξέρετε, στην Τουρκία επίκυνται εκλογές τον Ιούνιο. Ως εκ τούτου, θέλω να τονίσω ότι μονάχ, όχι μόνο από την πλευρά της εισηγήτριας, αλλά γενικά από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εμείς πράττουμε ό,τι είναι δυνατό για να εξασφαλίσουμε την ισορροπία αυτής της έκθεσης. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο για τα θέματα αυτά αφήρασα, ε, την τροπολογία 250. Και γι' αυτό θέλω να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να εξατάσουν και πάλι στις τροπο, τροπολογίες 6, 7, 12 και 13 καθώς και την 313 σε ό,τι αφορά την ικανότητα ενσωμάτωσης Και η 313 αφορά επίσης την ε, εισδοχή της Τουρκίας και την ικανότητα ενσωμάτωσης. Θέλω να σας υπογραμμίσω και πάλι ότι στις αιτιολογικές ε, σκέψεις α, β και γ ο στόχος μας είναι να αντανακλάται η θετική μας αντιμετώπιση. Και ελπίζω θα λάβετε υπόψη το γεγονός ότι έχει αποσυρθεί η τροπολογία 250 και να λάβετε επίση τι τροπολογίε 6, 7 <clears throat> και τα λοιπά ω 313 και να μην τις καταψηφίσετε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, αν δεν τις υποστηρίζετε. Ευχαριστούμε λοιπόν. Ο κύριος Χάουιτ. Δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση, απλώς διαδικαστικά θέλω να πω το εξής επειδή το ΕΛΚ αποσύρει την τροπολογία 250 ναι ναι να ελέγξω μια στιγμή επειδή έχει αποσύρει το ΕΛΚ την 250 εμείς θα αποσύρουμε την 6 και αν οι πράσινοι δεν αποσύρουν τη δική του τροπολογία θα την, θα την καταψηφίσουμε. Αυτή ήταν και η συμφωνία που κάναμε με την ε, εισηγήτρια για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες συμβασμού που με μεγάλη δυσκολία επιτύχαμε. Ο κύριος Μπρόκ θέλει να λάβει το λόγο. Ζήτησε προηγουμένως το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την κυρία Όμεν Ρόιτεν για την πρόταση που υπέβαλε. Βλέπω ότι και ο κύριος Χάουιτ ε, μετακινήθηκε προς μια σωστή κατεύθυνση σε ένα σημείο, αλλά δεν νομίζω ότι ε, υιοθετεί ολόκληρη την πρόταση της κυρίας Όμεν Ρόιτεν και αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολία που στην Ολομέλεια θα οδηγήσει σε αντιπαράθεση σε ένα σημαντικό θέμα. Και δεν ξέρω αν αυτό ε, θα ανοίξει τις δυνατότητες που έχουμε δηλαδή υπέρ της ένταξης της Τουρκίας θα πρέπει να, λάβουμε, να λάβουν υπόψη τους ότι έτσι ε, περιορίζονται οι δυνατότητες για κάτι τέτοιο στο μέλλον όχι μόνο στα πλαίσια του Κοινοβουλίου αλλά και για τις περαιτέρω ε, διαπραγματεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, Ας σε αυτά που ελέγχθησαν, οι έξι αποσύρεται, οι άλλες τροπολογίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Η εισηγήτρια παραμένει πιστή στην απόφασή της να αποσύρει τη 250. Ακόμα και αν δεν έγινε η συνολική αυτή ε, απόσυση τροπολογιών όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ των Ρωμανών. Η κυρία Ομεν Um, Αν μπορώ να ξαναγυρίσω στην προηγούμενη συμφωνία που είχαμε κάνει, που είχαμε ως πολιτικές ομάδες. Αν δεν τηρείται η συμφωνία, εμείς δεν μπορούμε να αποσύρουμε τη 250. Κοιτάξτε, λέει ο κύριος Χάουιτ. Θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των ομάδων και των εισηγητών. Εγώ σέβομαι τους κανόνες του Κοινοβουλίου και εάν εμείς κάνουμε κάτι καλή την πίστη σε ένα θέμα που ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο και πόσο ευαίσθητο είναι και στις πολιτικές ομάδες στο εσωτερικό τους αλλά και για το σύνολο του Κοινοβουλίου βλέπω ότι ο κύριος Μπρόκ έχει μια διαφορετική άποψη για την τροπολογία που αφορά την ικανότητα ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε είναι να στρεβλώνουμε τις συμφωνίες που έχουν γίνει σε συμβαστικό επίπεδο μεταξύ των ομάδων. Οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν χθε σε συμβαστικό επίπεδο για τις τροπολογίες 250, 6 και 7 και όχι τις άλλες τροπολογίες που έχει φέρει τελευταία στιγμή η κυρία Ομεν Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αλλάξει νόμοι τελευταία στιγμή. Αλλά μην δίνετε λανθασμένη εντύπωση για αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των ομάδων. Αν προσπαθούμε να έχουμε συνένεση, τότε, εάν θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή πλειοψηφία και να στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα προς την Τουρκία, τέτοιου είδους τακτικές τελευταία στιγμή δεν ωφελούν και δεν βοηθούν. Ο κύριος Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε, η ικανότητα ενσωμάτωσης ολοκλήρωσης ε, της Ένωσης και της Τουρκίας στην Ένωση θα αποφασιστεί από το Κοινοβούλιο. Εάν οι σοσιαλιστές θέλουν να μην αναφέρεται αυτό ως προϋπόθεση για την ένταξη της Τουρκίας, αυτό αποτελεί θέμα δημόσιας συζήτησης που την αποδέχομαι. Γι' αυτό δεν αποσύρθηκε 250. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι δυσκολεύεται αυτή η προσπάθεια εξέβρεση στην τελευταία στιγμή, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε και να δούμε τι θα γίνει στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι εμείς αποφασίσαμε τη θέση αυτή ε, ενώ για την ε, ικανότητα ολοκλήρωσης ενσωμάτωσης, ενώ οι σοσιαλιστές ε, υπαναχωρούν σε σχέση με τη συμφωνία. Η κυρία Όμεν πάντοτε τηρώ τις υποσχέσεις μου, αλλά χθες είπα στους συναδέλφους ότι οι τροπολογίες 11 και 13 είναι μεγάλη σημασία για μας. Αυτό είναι ένα. Δεύτερον, χθες το βράδυ δεν μπόρεσα να αποσύρω την 250 τροπολογία γιατί ο προτείνων, ο καταθέστης στην τροπολογία δεν συμφώνησε. Με, η κυρία Φλάστο δεν ε, συμφώνησε, δεν, μπορώ, μπόρεσα να τη βρω και οι 12 και 13 ψηφίστηκαν υπέρ. Και χθε είπα στους σοσιαλιστές συναδέλφους ότι το ΕΛΚ θα καταψηφίσει την 250. Αν υπάρχει κάποιος λοιπόν στο Κοινοβούλιο που μου λέει ότι δεν τηρώ τις υποσχέσεις μου και τις συμφωνίες, αυτό δεν αληθεύει. Εγώ ήθελα να κάνουμε μια συμφωνία σε βάθος. Ο κύριος Μποντής, μετά ο κύριος Χάουιτ, εδώ θα κλείσουμε. Ναι κύριε Πρόεδρε, η κυρία Βλαστό είναι αυτή η οποία κατά την τροπολογία 250 και η οποία δεν είναι παρούσα σήμερα το πρωί. Μου είπε μέσω του συνεργάτη της ότι μετά από την συνεννόησή της μαζί με την κυρία Όμεν Όμεν-Ρόιτεν θα αποσύρει πράγματι την τροπολογία 250. Χάουιτ, Μέσα στο πνεύμα αυτό του να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε καλές σχέσεις μεταξύ των κομμάτων θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Όμεν Ρόιτεν αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι κάνει μια διαφορετική προσφορά σήμερα το πρωί διαφορετική από αυτή που είπαμε χθες. Εμείς θα παραμείνουμε πιστοί στη συμφωνία αν δεν αποσύρουν τη 250 θα υπερψηφίσουμε την 6 και την 7. Το λέω σαφώς στον κύριο Μπρόκ και στην κυρία Όιμεν Ρόιτεν ότι θα επανέλθουμε και πάλι στην ψηφοφορία της Ολομέλης γιατί θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί. Αλλά αυτό το οποίο ελέγχθη νομίζω ότι καλύπτει την ε, ε, ανησυχία μου για μια παρουσίαση των πραγμάτων που δεν ήταν απόλυτα επακριβή. Ωραία, λέει ο πρόεδρο. Με τι διευκρινήσει αυτέ. μπορούμε να ψηφίσουμε. Αποσύρθηκε λοιπόν η 2.50 εφόσον δεν αποσύρονται οι υπόλοιπε. Εν πάση περιπτώσει τώρα θα ψηφίσουμε κατά περίπτωση όλες τις τροπολογίες. Θα ξεκινήσουμε με την τροπολογία 23. Ψήφι υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 22 υπέρ κατά απόχε απορρίπτεται 24 ψήφι υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 25 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 26 υπέρ κατά απόχες δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην 36 τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Η υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50. Όχι. 54. Όχι. Πάμε. να υπήρξε λάθος. Πάμε κατευθείαν στην 57 με χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της 57. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ θα λέγω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε έλεγχο. Ξεκινάει η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 36 υπέρ, 33 κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τη 57. <clears throat> Ψήφι υπέρ. Κατά. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είναι. Α ελέγξουμε όμω και εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα τη 57. Κάποιοι δεν ψηφίσουν πάντα, αλλά κλείνω την ψηφοφορία παρόλα αυτά. 35 υπέρ, 32 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 ψήφι <clears throat> υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ Θέλετε έλεγχο στην 68. Άρχεται η ψηφοφορία για την 68. Πέρας της ψηφοφορίας για την 68. 34-35 για μία μόνο ψήφο απορρίπτεται. 69 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 71 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, αλλά δεν είμαστε σίγουροι εδώ. Και κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 71. Άρχεται η ψηφοφορία για την 71. Κλείνει. 21 υπέρ 49 κατά. Ήταν σαφές, δεν είδα τα χέρια σας. Εν πάση περιπτώσει απορρίπτεται. 74 υπέρ. 74 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 Εντάξει, ηλεκτρονικό έλεγχο για την 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, chiusa la votazione. ψηφοφοριας ψηφοφορίας. 30-40 εγκρίνεται. Συμβαστή τροπολογία 6, ψήφι υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. 76 ψήφι υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. 77 υπέρ, Κατά. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται, αλλά ας είμαστε σίγουροι, <clears throat> κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για την 77. Πέρας. 36 υπέρ, 33 κατά εγκρίνεται. 78 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 85 ψήφι υπέρ κατά απόχες δεν είναι σαφές 85 ηλεκτρονική ψηφοφορία Έχουμε ένα σφάλμα στη διαδικασία ψηφοφορίας. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε την 85. Γιατί έχουμε εγκρίνει την 78. Πάμε στην 86 έχει αποσυρθεί όμως 87. Κάποιος θέλει να λάβει το λόγο. Η κυρία Φλότρα. Πράγματι, ελέγεται ότι αν η 78 εγκριθεί 85 εκπίπτει, αλλά πιστεύω ότι είναι συμβατές. Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε πράγματι την 85. If, if 78... Αν η 78 λέει κυρία Όμεν Ρόιτεν και διακόπτεται.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 Um, Κύριε Πρόεδρε, έχω κάποια νέα στοιχεία. Κατά την άποψή μου δεν ήταν συμβατή η 78 με την 85. Υπάρχουν κάποιες φήμες όμως στην Τουρκία που θα μπορούσαν να υπάρξουν περαιτέρω, ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν περαιτέρω έρευνε για, για τη δολοφονία του Χραντ Ντίνκ πριν από τέσσερα χρόνια. Οπότε α ψηφίσουμε. Και εγώ φυσικά υποστηρίζω αυτή την τροπολογία, εντάξει. Με αυτή τη διευκρίνηση είναι λίγο πιο, πιο εύκολο <clears throat> να είναι πιο εύκολο να θεωρήσουμε ότι είναι συμβατέ οι δύο αυτέ τροπολογίε. Ψηφίζουμε την 85 ψήφι υπέρ, λοιπόν. Ευχαριστώ κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Η 86 έχει αποσυρθεί λοιπόν, 87 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Ψήφι υπέρ. Κυρία Χάουιτ, για τη συμβαστική 10 υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος. Είπαμε ότι στη γραμμή 3 πρέπει να προσθεθούν οι λέξεις in this area, σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή, λυπούμε, θα εκφράζουμε τη λύπη μας ότι το 2010 δεν έχει γίνει καμία ε, μεταρρύθμιση σε, σε αυτό το χώρο, σε αυτή την περιοχή. Συμφωνεί. Αυτό ήταν απλώ διευκρίνηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αντιρρήσει να δεχτούμε αυτή τη διευκρίνηση από τον κύριο Χάουτ. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 10 με αυτή τη διευκρίνηση υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται 93 ψήφι υπέρ. Κατά αποχέ, απορρίπτεται. 94 έχει αποσυρθεί, 96 ψήφι υπέρ. Η 95 ναι, γιατί εκπίπτει αν, εγκρίνεται, αν εγκριθεί η 94. Η 94 έχει αποσυρθεί, οπότε πρέπει να ψηφίσουμε. Πρέπει να την ψηφίσουμε, λέει η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Ωραία, ωραία, ωραία, εντάξει. 95 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά δεν είναι σαφές για την 97 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 29 υπέρ 41 κατά απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 αποσύρθηκε, 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114. Ψήφι υπέρ. Μια στιγμή, μια στιγμή λέει ο πρόεδρος. Bene, 114 non si vota per... Δεν ψηφίζουμε την 114 γιατί είχε εγκριθεί η 50. Πάμε στη συμβαστική 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατόν λοιπόν υπέρ. Η κυριόμεν Ρόιτεν. Έχετε το λόγο. Αρχικά είχε γίνει ένα λάθος εδώ και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι καταψηφίσαμε την 119. Δεν την καταψηφίσαμε, κατέπεσε. Α, καλά, εντάξει, τότε λέει ο Όμεν Λοιπόν, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14. Ποιοι είναι υπέρ. Λοιπόν, συμβιβαστική 14. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επανερχόμαστε στο 122. 122 ψηφίζουμε. Chiusa la votazione. τη ψηφοφορία. 33 Λοιπόν, 33 κατά, 34 υπέρ δεκτή. Λοιπόν, συμβιβαστική 14. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. This is clear. Votazione elettronica. 130. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 130. Επαναλαμβάνει ο πρόεδρος για την 130 συμβιβα... ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Chiusa la votazione. 130. Chiusa la votazione. 37-32. Λοιπόν, απορρίπτεται 37 κατά 32 υπέρ. Εκατόν τριάντα ένα τριαντα Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 131. Ci sono sei colleghi che non Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 131 πέρα στις ψηφοφορίες. 48 κατά 18 υπέρ. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 145 υπέρ κατά τις 145 αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, οι 148 καταπίπτει, 150 ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Έχετε κουραστεί και δεν σηκώνετε τα χέρια σας και είναι δύσκολο να καταλάβω. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την 152 ηλεκτρονικά. Τέλος. 32 κατά 36 υπέρ. Δεκτή. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έχει αποσυρθεί 154, 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν μπορώ να καταλάβω πάλι. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 155 ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας 31 κατά 37 υπέρ δεκτή. 157 δεν την ψηφίζουμε. Η 158 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν είμαι σίγουρος όμως, την 161 την ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. 40 κατά 29 υπέρ απορρίπτεται. 162 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 170. Επανερχόμεθα στην 170. Ψηφίζουμε. Chiudiamo la votazione. 32 a 37. Λοιπόν, 32 κατά 37 υπέρ δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την 171 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έχει αποσυρθεί 175. 174 μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είδατε σας πρόλαβα κύριε Χάουιτ. Ξέρω τι θέλατε. Πριν από σας για σας. Α, εδώ έχουμε ένα επιπλέον σοσιαλιστή που θέλει να ψηφίσει. Λοιπόν, ένας από εσά δεν πρέπει, πρέπει να βγάλει την κάρτα. Chiusa la 39 no. Λοιπόν, 39 κατά, 25 υπέρ απορρίπτεται. 175 αποσύρθηκε, 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 181 τώρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. «183 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 184 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 191 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα υπέρ μου φαίνεται υπέρ, εν πάση περιπτώσει, εν περιπτώσει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 194. Ψηφίζουμε. Τέλος. 26 κατά 38 υπέρ γίνεται δεκτή 194. Τώρα όμως μου είπαν ότι πρέπει να πάμε πίσω και να ψηφίσουμε την 189 και την 191 γιατί είναι συμβατές με την 19 συμβιβαστική. Ψηφίζουμε την 189 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 190 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 194 τώρα υπέρ Α, όχι, την ψηφίσαμε ήδη την 194. 197 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν μπορώ να καταλάβω το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 197 παρακαλώ. 197. Chiusa la votazione sul 197. Λοιπόν, 51 υπέρ, 14 κατά. Τώρα, 198 υπέρ. Για την 198 υπέρ, κατά. Αποχές δεκτή. 199 υπέρ. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 198. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. «29 κατά, 38 υπέρ, δεκτή». Η 199 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. τα συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην 2.14 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται, έχει αποσυρθεί η 2.15, έχει αποσυρθεί η 207. Ψηφίζουμε την 200, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 205, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 207 αποσύρθηκε. Περνάμε στην 203. Τώρα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 211 υπέρ. Α, θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 203. Chiusa la votazione. Τέλος της ψηφοφορίας. 52 κατά, 14 υπέρ απορρίπτεται. Λοιπόν, 211 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 219 Λοιπόν την 218 την απορρίψαμε οπότε ψηφίζουμε την 217 μάλλον πρώτα 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 222 έχει ζητηθεί Chiusa la votazione elettronica. Λοιπόν, 45 κατά 21 υπέρ. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές Απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 230 ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. 31 κατά 30 υπέρ απερίφθη. Λοιπόν, η 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 233 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 234 υπέρ. 34 λοιπόν. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 235 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 236 υπέρ κατά αποχές δεκτή καταπίπτει 237 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 240 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 2.41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 246 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 247 υπέρ έχει αποσυρθεί μάλλον η 247 ψηφίζουμε την 248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 249 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τέλος φτάνουμε στο μυθικό 2.50. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. Α, α, το αποσύρατε. Θέλετε το λόγο, κυρία Όμεν Ρόιτεν. Κύριε Πρόεδρε, τη 250 είχα πει προηγουμένως ότι την αποσύρω ότι αυτή ήταν η πρόθεσή μας εφόσον οι σοσιαλιστές θα άλλαζαν την άποψή τους για την 12 και την 13 που αφορά την ε, δυνατότητα ενσωμάτωσης. Την έχουμε αποσύρει επομένω στη 250. Αλλά να το έχετε υπόψη σας αυτό όταν ψηφίσουμε τη 12, 13 και 413 και ας έχουν σοσιαλιστές το, μυαλό, το νου τους για το τι θα ψηφίσουν. Ο κύριος Χάουιτ. θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά ότι κατεγράφει αυτή η τροπολογία και δεν ψηφιστεί, γιατί εμείς θα ακολουθήσουμε τη συμβαστική λύση που δεχτήκαμε χθε το βράδυ, κύριε Πρόεδρε. Ας είμαστε σαφείς, λέει η κυρία Ομιλόντερ. Έχουμε μια νέα συμφωνία. Δεν συμφώνησα χθε το βράδυ να την αποσύρω, γιατί δεν είχα την άδεια της ομάδας μου. Σαν χειρονομία καλή θέληση την αποσύρω. Μετά από συνομιλία με την κυρία Βλαστό, αλλά θέλω και εσείς να τηρήσετε τη φόρμουλα στην οποία καταλήξαμε για τις άλλες τροπολογίες. Σας ζητώ και πάλι να αποσύρετε ή τουλάχιστον να καταψηφίσετε την 13, 14 και 413. Ωραία κατάλαβαν ποια είναι η θέση σα. Εγώ θέλω να ξέρω, όλοι μάλλον θέλουμε να το ξέρουμε αυτό, αν η συγγήτρια έχει πράγματι ούτω ή άλλω αποσύρει την 250 ή αν θέλει να την αποσύρει μόνο αν οι σοσιαλιστές αποσύρουν τη 12 και τη 13. Σας ρωτώ λοιπόν κυρία Όμεν αυτήν την ε, διευκρίνηση. Την αποσύρετε ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση ζητάτε να αποσυρθεί 12 και 13, αλλά αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση σαν καλή χειρονομία Καλή θέληση είναι χωρίς όρους η απόσυρση τη 250, αλλά τρέφω την ελπίδα ότι και η άλλη πλευρά θα δείξει θετικό πνεύμα. Ωραία. 250 αποσύρεται, 251 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.52 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 256 υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται 257 έχει αποσυρθεί 258 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 259 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 260 δεν την ψηφίζουμε 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 262 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 263 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές δεν Δεύτερο τμήμα της 263 με ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 32 υπέρ, 32, 36 κατά απορρίπτεται. 2,64 <clears throat> υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23 ψήφι υπέρ. 21 συγγνώμη. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.66 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.68 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.71 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε. Ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 276 azione. E eh, non, non si Chiusa la votazione. 31 υπέρ, 37 κατά απορρίπτεται πράγματι. 2,77 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές, όπως και οι προηγούμενοι. Απορρίπτεται. 2,78 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2.79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 282 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 22 <clears throat> ψήφι υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.84. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.85. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.90. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.91. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 291 ηλεκτρονικά. Σε Πέντε συνάδελφοι δεν ψηφίζουν, παρόλα αυτά κλείνουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία. 21 υπέρ 41 κατά απορρίπτεται. 2.92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.96 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 298 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 299 εκπίπτει 300 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 303 ψηφίσμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 305 ψήφι υπέρ 304 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. Άρχεται ψηφοφορία. Για την 304. Πέρας. 51 κατά, 17 υπέρ. Απορρίπτεται. 405. ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 406. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 307 υπέρ κατά αποχές από 308 υπέρ κατά αποχές από 309 υπέρ Λοιπόν, 308 ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. 9 δεν ψηφίσανε ακόμα. Πέντε. Δεν έχετε πιει καφέ ακόμα, μάλλον. Κάποιοι συνάδελφοι κοιμούνται, υπνώτουν. 16 υπέρ, 50 κατά, απέριπτε. 309 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτε. 310 υπέρ. κατά. Αποχές απορρίπτε. 311 και 312 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 313 υπέρ κατά δεν, δεν είναι σαφές ψηφοφορία ηλεκτρονική για 313 Era ένα Μία από τις επίμαχες τροπολογίες ήταν αυτέ που αναφερόταν στη συμφωνία των πολιτικών κομμάτων. Ε, ε, Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Πέρα τη ηλεκτρονική ψηφοφορία. 25 υπέρ, 37 κατά. Απορρίπτεται. 3-14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ την έχουμε αποσύρει, λέει ο κύριο ε, Χάουιτ. Πολύ ωραία. 8. Υπέρ, κατά, απόχέ. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ, κατά, απόχέ. Ε, απορρίπτεται. 10. Υπέρ, κατά, απόχέ, Απορρίπτεται. 11. Υπέρ, κατά, απόχέ, Απορρίπτεται. 12. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 ψηφίσμα ψήφι υπέρ κατά δεν είναι σαφές 14 ηλεκτρονικά Έξι συνάδελφοι δεν έχουν πιει καφέ και δεν ψηφίζουν. E Πέρασε. 47 κατά, 19 υπέρ, απορρίπτεται. 15 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 και 21 έχουν αποσυρθεί 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται εκπίπτει 3 πάμε στην 4 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται η ψηφοφορία Αν θέλετε να με ακούσετε για μια ακόμα φορά. Νομίζω έχουμε ξαναγυρίσει σε αυτά τα οποία ήταν το αντικείμενο της συμβαστικής ε, ε θέσης μας και τώρα χαίρομαι που έχουν μάθει οι σοσιαλιστές ότι είναι πολύ χρήσιμο να τηρούμε τις ε, συμφωνίες μα και είναι μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι μαζί σα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Όμεν πριν από την τελική ψηφοφορία και σας συγχαίρω και εγώ. Κλείνουμε την ψηφοφορία ενδιαμέσως με πέντε ψήφους κατά και τρεις αποχές 51 υπέρ έχει εγκριθεί συγχαρητήρια κυρία Όμεν και Ρόιτεν. Κύριε Ομπιόλς, εδώ και πολλά χρόνια έχω μάθει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις συμβιβαστικές, τροπολο... θέσεις και επίσης έμαθα ότι πρέπει να μαθαίνει κανείς να λέει και την αλήθεια για τις συμβαστικές αυτές θέσεις. Ο χθεσινός συμβιβασμός ήταν αυτός ακριβώς που τηρήσαμε εμείς. Θα ήθελα να καταγραφεί αυτά στα πρακτικά και φυσικά δεν δέχομαι από κανένα όσο και να τον εκτιμώ ούτε και από την κυρία Όμεν Ρόιτεν να μου δίνει μαθήματα για το αν πρέπει να σεβόμαστε να μην σεβόμαστε τους συμβιβασμούς στους οποίους προβαίνουμε. Καλώς. Παραχωρώ λοιπόν την Προεδρία στον κύριο Μποντίση για τη συνέχεια των εργασιών και σας ευχαριστώ. Γεια σας. vote pareil. Euh, nous poursuivons la séance. Point sur euh, la résolution concernant. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στην συζήτηση για την Φιρόμ. η κατάσταση στη χώρα αυτή ήταν σχετικά ανησυχητική μετά από μια απόφαση των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης να σαμποτάρουν τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τάλερ για να μας παρουσιάσει τα βασικά σημεία του ψηφίσματός του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου μετά από την όλος ενδιαφέρουσα ψηφοφορία για ένα υποψήφιο κράτος, την Τουρκία και την Κροατία, σήμερα συζητούμε για την πρόταση ψηφίσματος για το επόμενο ε, μελλοντικό μέλος στην πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας, την ΦΥΡΟΜΑ που ε, εντάσσεται σε καλή συντροφιά, γιατί θα μιλήσουμε για το Ισλάμ. Αν η πολιτική είναι και συμβολική, νομίζω ότι ε, είναι θετικό το γεγονός ότι τα σημερινά υποψήφια υποσυζήτηση μέλη μπορούν να ε, προχωρήσουν παράλληλα. Συζητούμε το ψήφισμα μια ημέρα κατά την οποία ιδρύεται μια σχέση φιλίας με τη χώρα αυτή. Έχει περάσει ένας χρόνος από το προηγούμενο ψήφισμά μας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και τώρα θα ήθελα να παρουσιάσω ορισμένα κύρια σημεία του τωρινού ψηφίσματος για την ΦΥΡΟΜ. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι η πρόταση ψηφίσματος προτείνει η χώρα Φιρόμ να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις ενταξιακές. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Είναι το κύριο μήνυμα του ψηφίσματος. Η Μακεδονία εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων. Άλλωστε αυτό το επιβεβαίωσε πριν από λίγους μήνες η έκθεση της Κομισιόν και η πρόταση ψηφίσματος προτείνει την έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών. Ε, λυπούμεθα διότι ακόμη δεν άρχισε το Συμβούλιο της Διαπραγματεύσης και προτείνουμε να προχωρήσει ε, στην σχετική απόφαση το Συμβούλιο. Όπως είπε ήδη ο Πρόεδρος, το ψήφισμα εκφράζει ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ΦΥΡΟΜ. Πρόκειται για τρεις προβληματικούς τομείς. Πρώτον, πολιτικός διάλογος στη χώρα ή καλύτερα η έλλειψη του διαλόγου αυτού που το τελευταίο διάστημα οδήγησε σε εμποϊκοτάστηση του κοινοβουλευτικού έργου από μια μεγάλη πλειοψηφία των αντιπολιτευομένων κομμάτων. Ένας άλλος προβληματικός τομέας είναι η δικαιοσύνη ή καλύτερα ή το θέμα της ανεξαρτησίας. Πρόκειται για την εξάρτηση της δικαιοσύνης εδώ. Τρίτον, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ή η έλλειψή τους και πάλι, ιδιαίτερα των ΜΜΕ που ασκούν κριτική. Το ψήφισμα εκφράζει έπαινο για το έργο του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια, ο οποίος ε, στην ε, πολύχρονη θητεία του επετέλεσε εξαιρετικό έργο. Είναι ο πρέσβης ε, Ντεφορέ, ο οποίος και τα Σαββατοκύριακα εργαζόταν για πρόοδο. Επίσης, είναι ε, ενδιαφέρον το γεγονό ότι και εκείνος ε, υπέστη προσωπικά επιθέσεις όπως και άλλοι εκπρόσωποι της Ένωσης και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή δεν είναι ε, σωστή συμπεριφορά. Στον τομέα του τύπου των ΜΜΕ υπάρχουν κάποια προβλήματα που κλιμακώθηκαν πρόσφατα με το τηλεοπτικό σταθμό Α1 και με βάση τις αντικειμενικές μετρήσεις είναι ο πλέον σημαντικός σταθμός σε ό,τι αφορά την επιρροή που ασκεί. Αυτή τη βδομάδα ε, άνοιξαν ε, οι λογαριασμοί του Λουσταθμού. Αυτό είναι σημαντικό που δείχνει ίσως ότι ε, καταλαβαίνει τη σημασία αυτών των σταθμών το κράτος. Επίσης, πρόσφατα το Υπουργείο Εσωτερικών στην ιστοσελίδα του ε, ζητεί οι πολίτες να καταγγέλουν τα μία αντικειμενικά άρθρα του, του τύπου. Αυτό ακούγεται παράδοξο. Έγινε όμως. Και ελπίζω ότι η κυβέρνηση των Σκοπίων θα λάβει υπόψη της ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είναι το προσήκον όργανο για να κρίνει την αντικειμενικότητα ή μη των άρθρων του τύπου. Παρόλες τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις, τις επικρίσεις, αν θέλετε, στην εξέλιξη στα Σκόπια, θα ήθελα να πω ότι στο ψήφισμα καταγράφονται και θετικές εξελίξεις και μία κάποια πρόοδος στη χώρα αυτή. έχω καταγράψει και τα θετικά σχόλια. 11 είναι, τα μέτρησα. Είναι διψήφιο το νούμερο λοιπόν των θετικών σχολείων και βλέπουμε πάνω σε αυτή τη βάση σε ποια σημεία και σε ποιους τομείς επετέλεσε πρόοδο η ΦΥΡΟΜ. Είναι σημαντικό σε αυτό το ψήφισμα και σε άλλα να υποδεικνύουμε που χρειάζεται πρόοδος, που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειάζεται ε, περισσότερη πρόοδος, ε, βελτίωση. Καλό θα ήταν να υπάρχει και ένα εγχειρίδιο για τα θεσμικά όργανα, ούτω ώστε να επικεντρώνονται στους κρίσιμους τομείς. Η μάχη κατά της διαφθοράς είναι πολύ σημαντικός τομέας. Χαιρετίζουμε την πρόοδο σε αυτό το τομέα. Παράλληλα, επιθυμούμε όμως να τονίσουμε ότι χρειάζεται αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, αλλά και αμεροληψία, αντικειμενικότητα ε, στην κατήσχηση των νόμων κατά της διαφθοράς. Είναι σημαντικό να εξεταστούν ορισμένε περιπτώσεις, υποθέσεις καλύτερα και πιο εντατικά από άλλους. Ε, φέτος γιορτάζομαι τη δεκαετή επέτειο της Συμφωνίας της Αχρίδας που ε, συνέβαλε στη βελτίωση των σχέσεων και στα πλαίσια του κράτους παραμένει η συμφωνία πλαίσια της Αχρίδας ε, σημαντική και οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις μεταξύ Σκοπίων και Βρυξελών σχετικά με το πώς θα εορταστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επέτειος αυτή. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι οι εσωτερικές σχέσεις ε, εξελίσσονται, δηλαδή οι σχέσεις μέσα στη χώρα εξελίσσονται θετικά. Επίσης είναι σημαντικό να ε, αναφέρομαι και την περιφερειακή διάσταση των προβλημάτων. Εδώ εκφράζει έναν έπαινο το ψήφισμα για το σταθεροποιητικό ρόλο της χώρας στην περιοχή, τονίζει τη συνεργασία στις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα όμως τονίζει ότι οι κοινέ ε, θέσεις της σκέπα θα πρέπει να τηρούνται από τη ΦΥΡΟΜ και αναφέρει ιδιαίτερα και τη περίπτωση της Ζιμπάμπου που η κυβέρνηση προχώρησε κάπως υπερβολικά. Επιτρέψτε μου τέλος να απευθύνω έκκληση προς εμάς τους παρόντες. Στη χώρα αυτή θα πρέπει να δούμε τις εντάσεις που υπάρχουν μεταξύ των πολιτικών παραγόντων. Υπάρχει έλλειψη διαλόγου, εκφράζεται ανοιχτή εχθρότητα ε, μεταξύ των πολιτικών προσωπικότητων και η έκκληση που απευθύνω είναι εμείς ως Ευρωπαίοι Ευρωβουλευτές να προσπαθήσουμε να μην ε, πάρουμε ε, θέση υποστηρίζοντας τους ε, τοπικούς παράγοντες γιατί εμείς ε, δεν είμαστε υποψήφοι που θα κατέβουν στη Βοσνία, Αρζεγοβίνη ή και στην Φύρομα αν θέλετε. Είναι σημαντικό να τονίζουμε ότι εδώ δεν πρόκειται για καταστάσεις άσπρου μαύρου και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ε, δεν πρέπει να λαμβάνουμε θέση υπέρ κομμάτων. Πρόκειται για σύνθετη κοινωνία εδώ και θα έλεγα ότι η διαμόρφωση ενιαίων θέσεων από εμά συμβάλλουν στις θετικές εξελίξεις. Ε, περιμένω τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, τις τροπολογίες σας. Ελπίζω να μην είναι πάρα πολλέ, αλλά θα τις δούμε σοβαρά. Τα πράγματα εξελίσσονται, οι εξελίξεις τρέχουν, άρα πρέπει να ε, αναπροσαρμόσουμε στην επικαιρότητα κάποια θέματα. Εγώ με ενδιαφέρον θα ακούσω τις παρεμβάσεις και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα πρέπει ο χρόνος ομιλίας των ε, βουλευτών που θα ακολουθήσουν. Θυμίζω ότι οι σκιώδεις εισηγητές έχουν τρία λεπτά και οι υπόλοιποι που θα πάρουν το λόγο ενάμιση λεπτό. Για την ομάδα των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρία Νικολάη. Η έκθεση του κ. Τάλερ είναι ισορροπημένη έκθεση, χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα. Θα ήθελα να προσθέσω, αν θέλετε, τρία επιπλέον σημεία. Πρώτον, θεωρώ ότι η πρόταση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να ακουστεί επιτέλους από το Συμβούλιο. Η Μακεδονία, λέει η ομιλήτρια, έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου, αν και παραμένουν ακόμα προβλήματα. Νομίζω ότι πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει υπάρξει πρόοδο στην εφαρμογή της Συμφωνίας της Αχρίδας και ελπίζω τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην Αλβανία τελευταία να μην επηρεάσουν αυτά που συμβαίνουν στην γειτονική χώρα. Τα βήματα πρόοδου στον τομέα της δικαιοσύνης πρέπει να σημειωθούν. Ζητάμε από τα Σκόπια να κάνουν περαιτέρω βήματα προόδου στον τομέα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης για να αποφεύγονται οι πολιτικές πιέσεις στη δικαιοσύνη. Σχετικά με τη συμπεριφορά της πολιτικής τάξης θα πρέπει να εξευρωπαϊστεί θα πρέπει να βελτιωθεί και θα πρέπει να υπάρξει συνεχής διάλογος αδιάκοπτος ανάμεσα στους πολιτικούς σχηματισμούς της συγκεκριμένης χώρας. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω το θετικό στοιχείο της βελτίωσης των σχέσεων με τη Σερβία. Η κατάργηση ελέγχου διαβατηρίων είναι μια πολύ καλή νέα συμφωνία και η συμφωνία για την ενέργεια επίσης η οποία είναι συμβατή με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι θα κρίνουμε ότι η έκθεση είναι επικοδομητική και θα υπάρξει μια συμφωνία ευρύτερη γύρω από τη Μακεδονία, λέει η ομιλήτρια. Ο κύριος Μπρόκ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο τώρα. Δυστυχώς πρέπει να φύγω και ζητώ την κατανόηση των συναδέλφων γι' αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Τάλερ για την έκθεσή του. Πράγματι πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να έχουμε μία θέση όσο πιο πολύ γίνεται και έτσι να ενισχύσουμε την μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Μακεδονία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το κλασικό θέμα που υπάρχει σε όλα τα κράτη, όπως η διαφθορά, διοίκηση, δικαιοσύνη και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις εκεί. Τώρα, για τα ΜΜΕ θα ζητούσα να γίνει μια έρευνα συγκεκριμένη, γιατί έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένας ε, σταθμός ε, φιλοκυβερνητικός, ενώ οι υπόλοιποι είναι επικριτικοί. Ίσως λοιπόν δεν ε, πρέπει να ανησυχούμε πολύ. Καλύτερα όμως να ξαναδούμε την κατάσταση και μπορεί εδώ να μας βοηθήσει η γραμματεία να γίνει μια, μια μελέτη. Ένα θέμα θέλω να θίξω που μου είναι σημαντικό. Πράγματι, ο πολιτικός διάλογος θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η διαίρεση σε αυτά τα κράτη και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι οξίες δεν είναι θετικές για την ε, πρόοδο της χώρας. Υπάρχει όμως ένα θέμα ξεκάθαρο. Μπορεί κανείς να βλέπει επικριτικά τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, να έχει άλλη γνώμη για τα ΜΜΕ, άλλη γνώμη για τη δικαιοσύνη κλπ. Όμως δεν είναι δυνατόν να αποσύρεται κάποιος από το κοινοβούλιο. Αυτό είναι άλλο επίπεδο πια είναι άλλο πράγμα να συνεργάζεται κανείς ως αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα δημοκρατικό καθήκον. Δεν υπάρχει όμως καμία ε, νομιμοποίηση ε, στη διακοπή του κοινοβουλευτικού έργου. Είναι απαράδεκτο, επειδή δεν συγκεντρώνει κάποιος την πλειοψηφία, να αποσύρεται. Αυτό δεν είναι δυνατό να γίνεται και θα πρέπει να το τονίσουμε και για τις γειτονικέ χώρες. Επιστροφή στο Κοινοβούλιο λοιπόν, εκεί θα πρέπει να ε, εκφραστούν οι θέσεις και εκεί θα πρέπει να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Έτσι λειτουργεί στην Ευρώπη η Δημοκρατία. Η άσκηση πιέσεων ε, ως μέθοδο συγκεκριμένη, διότι αποχώρησε από το Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να συγχωρηθεί και να γίνει αποδεκτή. Ευχαριστώ. Κυρία Εμπρισάκη, τρία λεπτά σκιώδη εισηγήτρια είστε. Κάτι λέει ο κύριο Στάνο και εκτός μικροφώνου δεν ακούγεται. Εγώ δεν είμαι σκιώδη εισηγήτρια, λέει η κυρία Εμπρισάκης. Ο συνάδελφος Κουκάν είναι ο σκιώδη εισηγητή. Κύριε Κούκαν, θέλετε εσείς το λόγο ή κυρία Εμπρισάκης στη θέση του κύριου Κούκαν. Και εγώ θέλω να μιλήσω, αλλά μετά από τον κύριο Κούκαν. Αυτό είναι ο σκιώδη εισηγητής μου. Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστήσω τον Τζόραν Τάλερ που παρουσιάσε ένα σοβαρό έγγραφο που μπορεί να αποτελέσει καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις. Οι περαιτέρω συζητήσεις χρειάζονται. Συμφωνώ ε, για την ανάγκη να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία σύντομα. Στην προηγούμενη έκθεσή μας του 2010 για τη Μακεδονία είχαμε αναγνωρίσει στέρεη πρόοδο και ελπίζομαι ότι η χώρα θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Λυπούμε λοιπόν διότι οι εξελίξεις δεν ήταν τόσο θετικές όσο περιμέναμε. Με ανησυχούν οι πρόσφατες πολιτικές εντάσεις στη χώρα. Είναι σαφές ότι το μποικοτάρισμα του Κοινοβουλίου από την αντιπολίτευση δεν είναι τρόπος επίλυσης αυτών των εντάσεων. Οι πολιτικές αντιφάσεις και διαφορές πρέπει να στηριχθούν σε πολιτικό διάλογο μέσα από τα θεσμικά όργανα που συστάθηκαν για αυτό το σκοπό. Αλλιώς θα υπάρξει εμβάθυνση των διαφορών και στο τέλος θα ε, καταλήξουν σε αδιέξοδο. Επίσης είδα ότι πολλοί μιλήσατε για την ελευθερία των ΜΜΕ. Συμφωνώ ότι το θέμα θα πρέπει να το δούμε όπως του αξίζει στα πλαίσια της έκθεσης, ιδιαίτερα στα πλαίσια της, ε, των προβλημάτων γύρω από το σταθμό Α1 και κάποιες άλλες εφημερίδες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ολοκλήρωσης ενσωμάτωσης, το να κρατήσουμε ε, την Μακεδονία ε, εκτός διαπραγματεύσεων για ένα χρόνο ακόμα δεν θα βοηθήσει να βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα. Αντίθετα φοβάμαι ότι κατά πάσα πιθανότητα πέρα από τα πολιτικά προβλήματα θα προσθεθούν και εθνοτικές, εθνικιστικές εντάσεις. Η Μακεδονία θα πρέπει να έχει μια θετική ατζέντα για να επικεντρωθεί απάνω εκεί. Και αυτή είναι η ευρωπαϊκή ατζέντα. Ελπίζω λοιπόν ότι ε, θα λυθούν τα προβλήματα ε, έναρξης των διαπραγματεύσεων. Μια περαιτέρω παράταση μετά από τόσα χρόνια μόνο αρνητικά θα επιφέρει όχι μόνο στη Μακεδονία αλλά και σε άλλες χώρες της περιοχής. Τέλος, Νομίζω ότι εμείς ως πολιτικοί θα πρέπει εδώ να δώσουμε περισσότερο όραμα, μεγαλύτερο όραμα και προοπτική στην περιοχή. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις θετικές αλλαγές στην χώρα και να μην τους κρατάμε πίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Κορνέλησεν. Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ Ζόραν για την έκθεσή σου, η οποία θίγει πολλά και σημαντικά θέματα. Ε, χαίρομαι διότι το, όνομα του, το θέμα του ονόματος είναι στο τέλος της ε, έκθεσης γιατί υπάρχουν άλλα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια η πολιτική κατάσταση τώρα είναι στο προσκήνιο. Νομίζω ότι δεν είναι καλό σημείο το γεγονός ότι η Μακεδονία σε σχέση με πέρσι έχει πιο πολλά εσωτερικά παρά εξωτερικά προβλήματα. Τώρα, το μποϊκοτάρισμα του Κοινοβουλίου δημιούργη, ήταν ε, ε, θέμα που δημιούργησε κατακραυγή. Συζητήθηκε πολύ, είναι επιζήμια εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντικό εμείς να διατηρήσουμε ως Κοινοβούλιο την άμεροληψία μας. Βέβαια πιέζουν τα μέλη των πολιτικών οικογενειών μας να υποστηρίξουμε τη μία ή την άλλη πλευρά. Και εμείς ακόμα, οι πράσινοι, υφιστάμεθα πιέσεις, παρόλο που το αντίστοιχο κόμμα είναι πολύ μικρό θα πρέπει να παραμείνουμε αμερόληπτοι. Το μποϊκοτάρισμα δεν είναι απάντηση. Θα πρέ... Ούτε όμως το παιχνίδι πάνω ε, ε, εξουσίας από την κυβέρνηση. Ελπίζω λοιπόν ότι όλα τα κόμματα θα συμφωνήσουν. Έχω δει και κάποια ανακοινοθέντα στον τύπο που είναι κατά αυτών των καταστάσεων. Επίσης, δεν είναι τόσο θέμα του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ περισσότερο θέμα πολιτικής κουλτούρας που δεν ε, είναι σημαντικό μόνο εδώ, αλλά και γενικότερα στο πώς αντιμετωπίζονται οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, στο πώς απευθύνονται οι πολιτικοί στα ΜΜΕ για τους άλλους, για τους συναδέλφους τους, για τις μειονότητες, αλλά και τον επικεφαλής της, της αντιπροσωπείας της Ένωσης. Κάτι άλλο επίσης, η διαδικασία αποκέντρωσης αναφέρεται στην έκθεση αυτό από ό,τι κατάλαβα όμως από του ΟΤΑ, αν θέλετε, στην ε, Μακεδονία, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ε, τους αναθέτουν καθήκοντα, αλλά όχι και τους απαραίτητους πόρους για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα. Οπότε αυτό πρέπει να το πούμε. Η περιβαλλοντική πολιτική... Μίλησα στον Πρωθυπουργό Γκρουεύσκη το Δεκέμβριο. Δεν φαίνεται να ξέρει και πάρα πολύ καλά τι είναι η περιβαλλοντική πολιτική, γιατί μίλησε μόνο για μία μέρα όπου φυτεύουν τα δέντρα το χρόνο. Αυτό φαίνεται ότι είναι το πιο, πιο σημαντική πτυχή της περιβαλλοντικής πολιτικής στη Μακεδονία, οπότε αυτό λιγάκι να το σπρώξουμε. Και τέλος το θέμα του ονόματος με απασχολεί και με στενοχωρεί, γιατί μείναμε στα ίδια τα περσινά και δεν έχει επιτελεστεί πρόοδος εδώ. Ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάποιο μηχανισμό επίλυσης των προβλημάτων των διμερών. Όχι μόνο για αυτή την περίπτωση, αλλά και για περιπτώσεις που θα προκύψουν στο μέλλον μεταξύ χωρών ε, διεύρυνσης και χωρών διεύρυνσης και χωρών μελών της Ένωσης. Ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να αρχίσουν να σκέφτονται το ενδεχόμενο κάποιων τέτοιων μηχανισμών ε, επίλυσης λύσεων που αντίστοιχα θα ε, τίθενται σε εφαρμογή. Ευχαριστώ κύριε Στάνοκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα να συγχαρώ τον Ζόραν για το σχέδιο έκθεσής του. Αλλά το πρώτο σχόλιο μου είναι, ότι ξεχάσατε ότι και το Μαυροβούνιο είναι μια υποψήφια χώρα όταν αναφερθήκατε στην Τουρκία και τη Μακεδονία. Ξεχάσατε ότι και το Μαυροβούνιο είναι υποψήφια χώρα. Εάν δεν το θυμόσαστε, αν το ξεχάσατε, σας το υπενθυμίσω. Η έκθεσή σας είναι πολύ πλήρης, σας συγχαίρω Κατά την άποψή μου όμως και την άποψη της ομάδας μου, ίσως δίνει μια πολύ αρνητική αντιμετώπιση για μια μικρή χώρα που αγωνίζεται εναντίον του μποϊκοταρίσματος του μεγάλου γείτονά τη και φύση που αγωνίζεται και κατά των εσωτερικών διαμαχών. Ελπίζω ότι θα διατηρηθεί το περιεχόμενο της συμφωνίας της Αχρίδας παρά την πίεση που ασκείται και έχουμε υποβάλει τροπολογίες για να τονίσουμε ιδιαίτερα το θέμα της ε, ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, τα προβλήματα των ε, εξωτερικών επενδύσεων που δεν είναι μονάχα θέμα της Μακεδονίας αλλά και άλλων περιοχών που, άλλων χωρών που θέλουν να προσελκύσουν περισσότερες εξωτερικές επενδύσεις. Πιστεύω επίσης για αυτά που είπατε για το, τις επικρίσεις εναντίον του επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας του Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας μιλήσει με πολλούς Μακεδόνες πολιτικούς, φαίνεται ότι κράτησε μια κάπως κομματική θέση και έκανε σχόλια στα μέσα ενημέρωση σχεδόν για όλα τα θέματα τα οποία ήταν υποσυζήτηση στο Μακεδονικό Κοινοβούλιο. Φέρω τα σαν αντιβασιλέα λιγάκι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια σωστή αντιμετώπιση για ένα διπλωμάτη. Τα θέματα αυτά πρέπει να αφαιθούν στους εγχώριους πολιτικούς, δεν εναπόκειται στους διπλωματικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπησέρχονται σε τέτοια θέματα. Πιστεύω λοιπόν ότι εν μέρη τουλάχιστον οι καταγγελίες αυτές θα πρέπει να ευσταθούν. Ακόμα και αν δεν μου αρέσουν οι προσωπικέ επιθέσει, αλλά νομίζω ότι οι διπλωμάτε δεν θα πρέπει να εμπλέκονται εκτό αν είναι απαραίτητο σε τέτοιε εσωτερικέ ε, διαμάχε. Η έκθεση επίση καταδεικνύει και το έργο το οποίο έχει γίνει για να υποστηριχθεί η κοινότητα των Ρωμά και δεν δέχομαι τα σχόλιά σα για την εκστρατεία κατά των αμβλώσεων. Εγώ προσωπικά είμαι κατά τη άμβλωση. Αυτό είναι θέμα συνείδηση στη χώρα μα. Και ο καθένα μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Εσεί έχετε τι απόψει σα και εγώ τι δικέ μου. Αλλά αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εσωτερικό επίπεδο στη Μακεδονία και αυτοί οι οποίοι έχουν ισχυρά συναισθήματα στη χώρα αυτή, αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Αυτό δεν πρέπει να συγχαίεται με την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιρλανδία απαγορεύει την άμβλωση και το σεβόμαστε αυτό. Αν και η Μακεδονία θέλει να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, είναι δικό τη θέμα. Και αν αναφερόστε σε μια εκστρατεία δημόσια, εγώ μπορώ να αναφέρω και αυτέ που γίνονται κατά του καπνίσματο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι η έκθεση πρέπει να σταθεί στο θέμα αυτό τη εκστρατεία κατά τη άμβλωση και εγώ θα υποβάλω προτάσει, τροπολογίε για να διαγραφεί αυτή η μνήμα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, λέει ο η κυρία Κοπά λόγο. Πρόεδρε, ε, θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Ζόραν Τάλερ για την ειλικρινή και έντιμη ματιά στην κατάσταση στη γειτονική χώρα. Όπως επισημαίνει, ε, σε πολλά προβλήματα αντί για, πρόεδρο, ε, πρόοδο είχαμε οπισθοδρόμηση. Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης πλήττεται, ο πολιτικός διάλογος είναι ανύπαρκτος με το μποϊκοτάζ της Βουλής από την αντιπολίτευση πράγμα που όπως επεσήμεναν πολλοί συνάδελφοι δεν συνάδει με τις αρχές ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος ε, δεν προχωράει καλά δεν στηρίζεται η αξιοκρατία και η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. σε όλα αυτά η κυβέρνηση του κυρίου γκρούευσκι απαντά με φυγή προς τα μπρος και με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην αρχαιολαγνία μέσα από το project ε, σκόπια 2014 και να έρθω στο θέμα του ονόματος. είναι γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης το πρόβλημα με το όνομα δεν λύθηκε. σήμερα όμως κανείς δεν μπορεί σοβαρά να υποστηρίξει ότι για όλα τα κακά της χώρας φταίει η ελλάδα. αν το όνομα είχε λυθεί δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τελειώνουμε με τη διαφορά ε, για το όνομα. η ελλάδα έχει κάνει προτάσεις τις έχει καταθέσει. δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά αλλά η διαφορά πρέπει να πάψει να αποτελεί το άλοθη του κύριου γκρούευσκη στο να μην εκπληρώνει τα κριτήρια της κοπενχάγης στο να φημώνει τον τύπο και να μην προχωρά σε πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας της οχρίδας. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον Ζόραν Τάλερ για την θετική αντιμετώπιση που έχει δείξει σε σχέση με το θέμα αυτό και την ε, πάρα πολύ εμπεριστατωμένη του έκθεση. Είναι δύσκολο να έχουμε θετικά στοιχεία για αυτή τη χώρα γιατί είναι μια νέα χώρα και οι ηγέτες της είναι και αυτοί πολύ νέοι αλλά όταν πρόκειται για τη δεύτερη εντολή μιας πολιτικής ελίτ που βρίσκεται στην εξουχησία στη χώρα αυτή, θα πρέπει να σκεφτούμε και ποια είναι τα πράγματα τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει ώστε να μην έχει δοθεί ακόμα η ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Και θα πρέπει να σκεφτούμε τι μπορεί να βοηθήσει και όχι οι νέες ενέργειες οι οποίες θα χωρίσουν τον λαό αυτής της χώρας από την Ευρώπη. Έχει δημιουργηθεί ένα τείχος που έχει το όνομα Μέγας Αλέξανδρος που ουσιαστικά εμποδίζει τη χώρα αυτή να λειτουργήσει και στο εσωτερικό και τη χωρίζει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν μια έλλειψη εσωτερικού διαλόγου μέσα στη χώρα αυτή μεταξύ των εθνοτικών κοινοτήτων και φυσικά και με τους γείτονες της χώρας αυτής. Θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να κάνω μια έκκληση στην πολιτική εξουσία της χώρας αυτής να αλλάξουν την αντιμετώπιση τους γιατί αυτό θα βοηθήσει και ιδιαίτερα στην διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Και πρέπει και από τη δική μας πλευρά βέβαια να υπάρξουν θετικές αντιμετωπίσεις. Αν εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ε, ενσωμάτωση της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουμε θετικά μηνύματα και από αυτούς οι επιθέσεις κατά του πρώην εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, χώρα αυτή είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το επικροτώ. Μπορεί κανείς να έχει υποπέσει σε σφάλματα, αλλά ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει καλή την πίστη πιστεύω. Δεν μπορεί να την κάνει τέτοιων ε, επιθέσεων. Θα πρέπει καταρχήν να κοιτάξουν στον καθρέφτη το πρόσωπό του στον καθρέφτη πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία και μετά να επιτίθεται κάτι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κ. Κόβατσεκ. Σα ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Ζάλερ για το έργο του σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματο. Ξέρουμε ότι όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τα Δυτικά Βαλκάνια είναι πολυδιάστατα και πολιτικά ευαίσθητα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να συνεχίσουμε να υποστηρί... παρά να υποστηρίζουμε τη μεταρρύθμιση στην Μακεδονία αλλά δεν πρέπει να αφιστούμε επικρίσεων σε θέματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι αυτά που έχουν γίνει με τα μέσα ενημέρωσης είναι πρόβλημα και επίσης τα προβλήματα με την μεγαλύτερη ιδιωτική τηλεόραση στην Α1 είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Και επίσης ανησυχώ για τις διακρίσεις που υφίστανται άτομα με βουλγαρική εθνοτική ταυτότητα. Και είναι πολλοί αυτοί στην ε, Μακεδονία. Δυστυχώ, τα άτομα αυτά πολλές φορές έχουν τύχει κακομεταχείρισης και έχουν υποστεί αυθαίρετε διακρίσεις, ακόμα και φυλάκιση και ε, έλλειψη πρόσβασης στην εργασία. Είναι πολύ αντικό να βλέπουμε να επανέρχεται η γλώσσα του μίσου στη μακεδονική κοινωνία που υποστηρίζεται πολλές φορές από του τοπικού ε, ιστορικούς. Όπως έχει λεχθεί, τα Βαλκάνια έχουν παραγάγει περισσότερη ιστορία από ό,τι έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν. Δεν πρέπει λοιπόν να αναμοχλεύουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, αλλά θα πρέπει αντίθετα οι πολίτε αυτή τη περιοχή να δουν ε, αντικειμενικά την ε, ιστορία τους και επίσης δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτού οι οποίοι είχαν εμπλακεί στο προηγούμενο κομμουνιστικό καθεστώ να δίνουν τον τόνο. Πρέπει η χώρα αυτή να σπάσει αυτό το δεσμό με το κομμουνιστικό παρελθόν και την ιδεολογική μονομερή ερμηνεία της ιστορίας. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν στη Μακεδονία, αν η Μακεδονία θέλει πράγματι να γίνει μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν ήθελα μια γενική παρατήρηση να κάνω. Νομίζω ότι με την έκθεση που συζητάμε σήμερα αδικείται ο λαός της ε, πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της ε, Μακεδονίας διότι όπως συνηθίζεται ζητάμε διάφορα πράγματα χωρίς να λέμε το πιο ουσιαστικό που θα έπρεπε να κάνει η Επιτροπή μας να κριτικάρει την Κομισιόν και το Συμβούλιο για την πολιτική της απέναντι στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και γενικά κύριε Πρόεδρε θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχουν εκθέσεις οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς ως αφετ να μην τοποθετούμαστε πάνω σε εκθέσεις των οργάνων αλλά να επιδιδούμαστε σε μια επιτρέψτε μου να πω έκθεση ιδεών όσον αφορά την κατάσταση σε μια τόσο σημαντική χώρα όπως είναι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεύτερο σοβαρό ζήτημα κύριε Πρόεδρε είναι ότι η κατάσταση που υπάρχει στη χώρα αυτή είναι προφανώς συνέπεια και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί πέρα, των οικονομικών και άλλων γενικότερων πολιτικών για τις οποίες δεν λέμε τσιμουδιά. Επίση, η έκθεση δεν λέει τίποτα για τι συνδικαλιστικέ ελευθερίε και τα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Μιλάει βέβαια για την ανεργία, αλλά γιατί γίνεται τις επιχειρήσει και αναφέρουμε και σε ελληνικέ επιχειρήσει, όπου στην ουσία δεν υπάρχουν συνδικαλιστικέ ελευθερίε, δεν γίνεται καμία συζήτηση. Επίση για το θέμα του ονόματο, θα ήθελα να πω ότι οι ελληνικέ επιχειρήσει που δραστηριούνται εκεί πέρα δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το όνομα, όπω και η γειτονική χώρα και τέλος να σημειώσω ότι η αναφορά που γίνεται στο σημείο 25 για ε, πολιτική ηγεσία εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίλυση του θέματος του ονόματος πρέπει να συμπληρωθεί πάνω σε ποια βάση θα γίνει η όποια διαμεσολάβηση, πολύ περισσότερο που η έκθεση δεν αναφέρεται καθόλου στις προσπάθειες που γίνονται από τον ε, ειδικό απεσταλμένο του ΟΕΕ για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Merci, monsieur. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Τάλερ για την έκθεσή του και επίσης την πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας για την πρόοδο την οποία έχει επιτύχει. Βέβαια υπάρχουν ακόμα εσωτερικές εντάσεις στη χώρα αυτή. Χαίρομαι που η έκθεση του κυρίου Τάλερ τονίζει ότι έχουν γίνει πρόοδοι και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Για ορισμένα θέματα όμως ίσως πρέπει να είμαστε σωστά, σωστά επικριτικοί, όχι υπερβολικά κριτικοί. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο φιλική αντιμετώπιση χωρίς να παραγνωρίσουμε και να αρνηθούμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει την φιλοδοξία να είναι υποψήφια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει παρετηθεί από τις φιλοδοξίες της λοιπόν και όπως είπε και ο εισηγητής θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα νέα στοιχεία στην έκθεση αυτή και ιδιαίτερα στην παράγραφο 11 είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι πρόσφατα έχει χαραχθεί μια νέα στρατηγική για τη δημόσια διοίκηση και επίσης στις παραγράφους 18 και 19 πρέπει να αναφερθούν οι προσπάθειες της κυβερνήσης σε σχέση με την κατάρτιση των νέων οι οποίοι ψάχνουν κάποια θέση απασχόλησης για πρώτη φορά. Δεν θα ήμουν λοιπόν τόσο σκληρός σε σχέση με τα θέματα των εξωτερικών επενδύσεων σε καιρό <clears throat> κρίσεων. Είναι δύσκολο να προσελκύσει κανείς εξωτερικές ε, επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το, τον αποκλεισμό κατά κάποιο τρόπο της, της ε, Πουδουγούμου, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Κούκαν, ότι εμείς θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα εσωτερικά θέματα της ε, Μακεδονίας και εμείς δεν έχουμε καμιά απολύτως αμφιβολία γι' αυτό ως κόμμα. Κύριε Μπρίζατζιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Τάλερ για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι το περιεχόμενο είναι ισορροπημένο. Σε ορισμένα σημεία ε, ίσως ε, θα τόνιζα τις προόδους πρώτα και μετά τους προβληματικούς τομείς. Ε, σχετικά μπορεί να υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Επίσης υπογραμμίζω αυτό που ανέφεραν κάποιοι προλαλήσαντες. Η πολιτική μάχη γίνεται στα σχετικά θεσμικά όργανα, όχι στο δρόμο. Είναι εντελώς απαράδεκτο ε, να εγκαταλείπει κανείς το κοινοβούλιο και μετά να επικρίνει ε, τη μη επίτευξη των στόχων που υποσχέθηκαν στους πολίτες. Μέσα στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να δίνεται η μάχη. Να επαναλάβω επίσης κάτι που το λέω εδώ και 5-6 χρόνια, γιατί πριν από ε, χρόνια ήμουν εισηγήτρια για τη χώρα αυτή. Θα πρέπει να ε, είμαστε προσεκτικοί τι μηνύματα αποστέλουμε προς τη χώρα. αν κάποιος τελειώσει, ε, περάσει τρία χρόνια χωρίς να επιτελέσει πρόοδο, τότε τι ε, περιμένουμε να ε, πιστέψουν οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Είναι όμως και θα πρέπει να τους δώσουμε το μήνυμα ότι όταν τελειώσουν με ένα θέμα μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Δεν μπορεί, συμφωνώ με τον κύριο Κούκαν, δεν μπορεί πια να περιμένει πολύ η χώρα αυτή μέχρι να της δοθεί το σήμα για τις προενταξιακές διαδικασίες. Ο κύριος Βόμποντα, ευχαριστώ. Να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στη χώρα. Τα εκλεγμένα κόμματα, όπως είπαν όλοι, πρέπει να έρθουν στο Κοινοβούλιο Ράμα, Μπερίσα, ε, και ε, αυτό εκφράζεται σαφώς στην ωραία έκθεση του κυρίου Τάλερ. Δεν χρειάζεται συζήτηση. Θέλω όμως ε, να αναφερθώ σε αυτό που είπε η συνάδελφος πριν από λίγο. Και εμείς θέλουμε η χώρα το ταχύτερο δυνατόν να πάει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η τωρινή κυβέρνηση θέτει το ένα μέτρο μετά το άλλο για να προκαλέσει τη γείτονα Ελλάδα. Εγώ δεν θέλω να ταχθούμε υπέρ, ή της, υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, δεν γίνεται. Αλλά δεν μπορώ, δηλαδή όταν ε, το, ε, συνεχίζουμε να λέμε ο Μέγας Αλέξανδρος το ένα, ο Μέγας Αλέξανδρος το άλλο, είναι πρόκληση. Δηλαδή συνεχώς σε μια προβληματική κατάσταση ε, δρώ προβοκατόρικα. Και προφανώς ε, ε, θα πρέπει στο Κοινοβούλιο να αρχίσει ένας πολιτικός διάλογος και ας φύγουν πια ε, από αυτό το στενό εθνικισμό και ας ανοίξουν προς την Ευρώπη. Αυτό νομίζω ότι όλους θα τους ωφελήσει και θα συμβάλλει και στο άνοιγμα των διαπραγματεύσεων και συζητήσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάλερ για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. δεν έχουμε πολύ χρόνο πια. Θα είμαι σύντομος, ευχαριστώ για την υποστήριξη αλλά και ε, την κριτική των συναδέλφων. Θα βελτιωθεί έτσι το κείμενο. Ε, ε, ε συγγνώμη που ξέχασα το Μαυροβούνιο που είναι υποψήφια χώρα πολύ σημαντική. Προσβλέπω στη συνέχιση της συζήτησης και την έγκριση του ψηφίσματος τον Απρίλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, στο θέμα του Ιράκ. Του Ιράκ είπα και του μέλλοντο των σχέσεων του Ιράκ με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σημεία 8 και 9 μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. όπω ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των προγραμμάτων και των εργαλείων συμβάλλει στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την πολιτική μετάβαση στο Ιράκ και την σταθεροποίηση του. <clears throat> Είναι λοιπόν Κάτι το οποίο ενισχύεται και με την πρόσφατη υπεογραφή μια συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία με την Ιρακινή κυβέρνηση. Είναι οι πρώτε συμβατικέ σχέσει που έχουμε πλέον με το Ιράκ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει θέση για αυτή τη συμφωνία επί τη βάση της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης. Ο κύριος Μάριο Μάουρο είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό και τον καλό να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε ήδη, στόχος αυτής της ανταλλαγής απόψεων, θέμα μάλλον, είναι η συμφωνία ανάμεσα στο Ιράκ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι για πρώτη φορά που υπογράφεται μια τέτοια συμφωνία. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει και μία πρόταση ψηφίσματος που να συνοδεύσει τη συμφωνία αυτή από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί να υπάρχει λοιπόν συνοδευτικό θα έλεγα ψήφισμα για τη συμφωνία που προβλέπεται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράκ. Για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει σχέση με το ότι το Ιράκ περνάει από μια πάρα πολύ ευαίσθητη φάση τουλάχιστον σχετικά με τις ευκαιρίες τις οποίες έχει και με την θέση την οποία θέλει να έχει στον αραβικό κόσμο, ο οποίος με τόσο απρόβλεπτο και εκπληκτικό τρόπο εξελίσσεται σε άλλες χώρες της περιοχής. Η χώρα αυτή, το Ιράκ, έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική θέση γεωγραφικά και το μέλλον της χώρας αυτής θα επηρεάσει άμεσα και το μέλλον των γειτονικών της χωρών. Ο ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Παράλληλα πιστεύω ότι στην κοινωνία των πολιτών στο Ιράκ τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχύσει την επιθυμία των πολιτών της χώρας αυτής να τους αντιμετωπίζουμε με εμπιστοσύνη. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να εκφραστεί με μία φωνή σχετικά με τις προοπτικές της δημοκρατικής εξέλιξης της χώρας αυτής. Πιστεύω λοιπόν στις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών του Ιράκ. Το Ιράκ δεν είναι μόνο το Ιράκ των βομβιστικών ενεργειών και των δολοφονιών και των ιδεολειπτικών και φιλετικών διαφορών. Αντίθετα, το Ιράκ περιλαμβάνει μια κοινωνία καταπιεσμένη, η οποία όμως έχει πάρα πολλές πολιτιστικές επιχειρηματικές δυνατότητες, έχει δυνατότητες επικοινωνίας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε ένα έγγραφο το οποίο να επιτρέψει στην κοινωνία του Ιράκ να δει την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια ευκαιρία και όχι σαν ένα διεθνές υποκείμενο σε εισαγωγικά το οποίο απλά συνάπτει εμπορικού τύπου συμφωνίες. Συνεπώς, πρέπει να υποστηρίξουμε τη συμφωνία αυτή με τη χώρα Ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και με τους συναδέλφους που έχουν αναλάβει σκιώδεις εισηγητές. Αυτή τη στιγμή περάσουμε σε περαιτέρω συζητήσεις και όχι μόνο εντός της Επιτροπής μας. Και εύχομαι επίσης να μπορέσω με όλους τους συναδέλφους να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ θέσει και κρίσεις τις οποίες προς στιγμή δεν έχω εντάξει στην πρότασή μου αλλά γύρω από αυτές είμαι απόλυτα δεκτικός. Τι εννοώ και στην έκθεση και στη συμφωνία δεν τίθεται το θέμα των ενεργειακών πόρων ή δεν τίθεται με δεσμευτικό τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε εμείς να εκφέρουμε μια άποψη γύρω από το θέμα της ενέργειας. Εγώ σαν παράδειγμα θα ήθελα να είμαστε ε, διαθέσιμοι να συζητήσουμε το θέμα της Αμερικανικών στρατευμάτων, όχι σαν αντικείμενο κριτικής του παρελθόντος, αλλά σαν σχολιασμό του Ιράκ του μέλλοντος, το οποίο είναι σε θέση να δρέψει τις ευκαιρίες που έχει μπροστά του. Συνεπώς, και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου θα αργήσει λίγο, νομίζω ότι έχουμε χρόνο να διοργανώσουμε και μία ακρόαση, τουλάχιστον μία, για να συναντήσουμε και το άλλο Ιράκ, το Ιράκ που δείχνει πόσο καλό είναι και πόσο έχει υπάρξει ανάκτηση δυναμισμού από την κοινωνία των πολιτών της χώρας. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι από πλευράς της υπηρετίας εξωτερικών ε, υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ε, διοριστεί ο νέος πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Έχουμε μια ακόμη ευκαιρία λοιπόν να συζητήσουμε να προχωρήσουμε σε λήψεις θέσεις θετικές σε σχέση με έναν στρατηγικό πάρτνερ, με μια κοινωνία 40 εκατομμυρίων πολιτών που περιμένουν από εμά να τους βοηθήσουμε. Όχι να τους πούμε μόνο ότι έχουμε υπογράψει μια συμφωνία, αλλά να τους καθοδηγήσουμε πολιτικά να στηρίξουμε το αίτημά τους για περισσότερη ελευθερία, δημοκρατία, ανάπτυξη και ευημερία είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα πιεστικό σαν αίτημα από όλα τα επίπεδα της Ιρακινής κοινωνίας. Πρόθεσή μου σε αυτή τη φάση είναι απλά να σας ακούσω, να κάνετε παρατηρήσεις και να μπορέσουμε έτσι στη συνέχιση της διαδικασίας να καταλήξουμε σε ένα κείμενο ιδιαίτερα παραγωγικό. Θυμίζω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 16η Φεβρουαρίου. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει ακόμα και ιστεροτέρα να επανέλθουμε στη συζήτηση ε, για το τι συμβαίνει στο Ιράκ σήμερα. Σας ευχαριστώ κυρία Κοπά, η οποία είναι σκιωδής για τους σοσιαλιστές. Τρία λεπτά. Merci, le Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μάουρο για την έκθεσή του δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και το οποίο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για μας και για τη σύνολη περιοχή. Είναι καλό μήνυμα το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να δεχτεί να αναβαθμίσει αυτή τη συμφωνία σε μια συμφωνία εταιρική σχέση. Ακόμα όμω δεν ξέρουμε γιατί καθυστερεί η υπογραφή αυτή τη συμφωνία και θα ήθελα να ακούσω από τα χείλη του Συμβουλίου τη Κομισιόν ποιο είναι ο λόγο για κάτι τέτοιο. Έχω επίση διαφορετικέ ε, πληροφορίε για την καταληκτική προθεσμία. Είπε η γραμματεία μας ότι και η προθεσμία για τι τροπολογίες θα αναβληθεί. Δεν ξέρω αν έχει περισσότερε πληροφορίε ο κ. Μάουρ για το θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν συγκρούμενε πληροφορίε. Η δημιουργία τη νέα κυβέρνηση δημιουργεί τη βάση για τη ριζοσπαστική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα αυτή να προωθεί στην εθνική συμφιλίωση σε μια κατακαιρματισμένη κοινωνία, να ενισχύσει την ασφάλεια και να προστατεύσει αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κ. Μαόρο έχει παρουσιάσει μια πλήρη έκθεση δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιθέσεις κατά των χριστιανικών μειονοτήτων στο Ιράκ, αλλά αφήνοντας κατά μέρο ίσως ορισμένα σημεία που είναι πολύ σημαντικά για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Εμείς πιστεύουμε ότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και τα ίδια προβλήματα όπως και οι άλλες εθνοτικές και θρησκευτικέ ομάδες στη χώρα αυτή, λόγω ακριβώς της κοινωνικής του κοινωνικού και κατακαιρματισμού, τη ένδυα, των προβλημάτων που σχετίζονται με την έλλειψη κράτου δικαίου κτλ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί του όμω και να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τα θέματα αυτά. Οχτώ μήνε μετά από τι εκλογέ, ο Αλμαλή κατάφερε να δημιουργήσει μια νέα κυβέρνηση συνασπισμού. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα πολλά θέματα τα οποία μένουν ακόμα εκκρεμή και κυρίως να μπορεί να επιτύχει το στόχο του να υπάρχει μια κρατική εξουσία σταθερή και ασφαλής, να έχει φιλικές σχέσεις με τους γείτονές της, να είναι μέσα στην διεθνή κοινότητα και να έχει κυρίως τη σταθερότητα. Μας ενδιαφέρει καταρχήν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου η κατάσταση είναι ακόμα ικτρή, έχει επαναφερθεί η θανατική ποινή και υπάρχουν καταγγελίες ότι υπάρχουν μυστικές φυλακές, φυλακές του Υπουργείου Εσωτερικών, ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά εγκρυπτό. Αυτό το αρνείται ο Αλ Αλμόλοκ, αλλά η Human Rights Watch στην έκθεσή της, την πρόσφατη, λέει ότι υπάρχουν πράγματι τέτοια κέντρα κράτηση. Αυτό είναι επίση θέμα ελευθερίας του τύπου, θέμα να σταματήσουν τα βασανιστήρια και κακομεταχείριση των κρατουμένων. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μνήμα στην κατάσταση των γυναικών. Όπω είναι σήμερα τα πράγματα, οι γυναίκε βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από την εποχή του Σαντάμ υπάρχει πολυγαμία, αγοράζονται οι γυναίκες για να τις παντρευτούν, δεν μπορούν να έχουν ένα διαβατήριο χωρίς την άδεια του συζύγου, όλα αυτά δείχνουν πόσο δύσκολο να είναι κανείς γυναίκα στο Ιράκ. Βάσει του συντάγματος το οποίο ενεκρίθη το 2005, υπάρχει ακόμα το θέμα του προσωπικού καθεστώτος, το οποίο βασίζεται στις παραδοσιακές σχέσεις. Επίσης μας ενδιαφέρει ότι όλες οι εθνοτικές και εθνικευτικές συνιστώσεις να ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Λόγω της δράσεως πολιτοφυλακών και ανταρτικών ομάδων που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι Αμερικανοί, εξακολουθεί να υπάρχει ανασφάλεια. Οι προτάσεις μας λοιπόν ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχω πολύ χρόνο, <clears throat> επομένως δεν θα πω περισσότερο, αλλά οι τροπολογίες μας θα ακολουθήσουν αυτή τη γενική κατεύθυνση, θα εργαστούμε περιεκτικά, δημοκρατικά, για ένα κράτος δικαίου το οποίο θα είναι υπέρ όλων των πολιτών και της περιοχής. Ευχαριστώ. Merci, euh, Kachin. Κύριος Κατσίν, για ε, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως σκιώδης εισηγητής Θέλω να ευχαριστήσω τον Μάριο Μάουρο για την εξαιρετική πρώτη φάση της έκθεσης. Είναι καλή βάση για να προχωρήσουμε. Το Ιράκ πρέπει να το προσέξουμε αλλά και να το βοηθήσουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι μακριά από μας το Ιράκ. Γι' αυτό τονίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την αντιπροσωπεία του να έχει φυσική παρουσία στο Ιράκ και εκεί να κάνει διάλογο με τις αρχές. Χαιρετίζω και την νομοδότηση του κυρίου Ταλαμπανή που είναι κατά της θανατικής ποινής και δεν θέλει να υπογράψει σχετικό διάταγμα παρά την επιθυμία της υπόλοιπης πολιτικής ελίτ. Η κατάσταση στο Ιράκ ε, ε, έχει γίνει θετικότερη, είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να χαιρετήσουμε την πρόοδο που συντελείται σε πολλούς τομείς. Το Ιρακινό Κουρδιστάν είναι τώρα ήσυχη, σταθερή και πολλά υποσχόμενη περιοχή όπου η χώρα είναι φυσιολογική, θα αρχίσουν ε, να ανοίγουν προξενία, η οικονομία ανθεί, οι υποδομές εξελίσσονται, η γεωργία επίσης και καθημερινά βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και προοδεύει το κράτος. Αν δεν πάμε στην Βαγδάτη, καλό είναι να πάμε στο Ερπίδιβιρ για να υποστηρίξουμε τις σταθεροποιητικές προσπάθειες που διευρύνονται από το Κουρδιστάν και αλλού. Δεύτερον, να τονίσω ότι οι προκλήσεις ε, όπως είδαμε στο Τίγρη στη, σε τρεις περιοχές δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε και να φέρουμε και εμείς από την Ευρώπη ειδήσει. Επίσης να καλέσω τον πρόεδρο Μαλίκη να σχηματίσει κυβέρνηση επιτέλους. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος όπως το Ιράκ χωρίς υπουργού σε σπουδαία χαρτοφυλάκια. δεν υπάρχει υπουργό εσωτερικών, υπουργό Άμυνα. Συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σήμερα στις Ιρακινές φυλακές. Θα πρέπει να δημιουργηθεί κράτος δικαίου. Γι' αυτό όλες οι αρμόδιες αρχές το ταχύτερο δυνατόν πρέπει να λειτουργήσουν και να αναλάβουν ενεργό δράση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός Μαλίκη ήδη ανακοίνωσε, και αυτό είναι θετικό, ότι δεν θα υποβάλει την επόμενη φορά υποψηφιότητα. Οι ταραχές στη Νότια Μεσόγειο έφτασαν και μέχρι το Ιράκ από ό,τι φαίνεται και ελπίζουμε ότι θα αντλήσουν σοβαρά διδάγματα και θα αρχίσει να λειτουργεί σύντομα η κυβέρνηση εκεί. Η κυρία Μπρέπολς, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ εξ ονόματος των Πρασίνων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Μάριο Μάουρο για το μέχρι δε έργο του. Εκτός αυτού νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι επιθυμεί να συνεργαστεί στενά με όλες τις πολιτικές ομάδες για να βελτιωθεί κι άλλο το ψήφισμα. Πολύ σύντομα για τις συστάσεις και τη συμφωνία συνεργασίας. Η συμφωνία είναι πολύ καλό βήμα προς μεγαλύτερη ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Κατά τις συνομιλίες που θα έχουμε τις την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες εβδομάδες με τον κύριο Μάουρο, θα πρέπει να επισέλθουμε και στην αιτιολογική έκθεση στο ψήφισμα. Τώρα, για το ψήφισμα καθ' αυτό. Οπωσδήποτε χρειάζεται ψήφισμα και εδώ επαναλαμβάνω τη συνάδελφο από τη σοσιαλιστική ομάδα εις ό,τι αφορά την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών γιατί μας είπε η γραμματεία ότι θα μας δώσει λίγο χρόνο παραπάνω. Ίσως λοιπόν μπορούμε αυτό κάπως στα γρήγορα να το συζητήσουμε. Κάποια σημεία τώρα που θα θέλαμε να τα φωτίσει το ψήφισμα περισσότερο. Πρώτον, το ζήτημα της θανατικής ποινής. Πολύ σύντομα γίνεται μία μνήα του Ταρίκα αλλά πιστεύουμε ότι το θέμα χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη παρά το γεγονός ότι το Ιράκ είναι μία από τις χώρες όπου επιβάλλονται οι περισσότερες θανατικές ε, καταδίκες στο ψήφισμα δεν λέει πολλά. Επίσης η αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα πρέπει να ε, παρουσιαστεί πιο καλά. Επίσης, αποπολιτικοποίηση ε, των ε, δυνάμεων ασφαλείας που θέλουμε και το ζήτημα της κακοποίησης κρατουμένων στις Ιρακινές φυλακές. Οι αμερικανικές πρακτικές κατά την περίοδο κατοχής στο Ιράκ πρέπει να αναφερθούν. Αλλά δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το παρελθόν. Εδώ ο κύριος Μάουρο έχει δίκιο. Θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Όμως, παρόλα αυτά, το θέμα πρέπει να το δούμε καλύτερα. Μετά, η ελευθερία του τύπου, των ΜΜΕ Ε, θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε αυτό το θέμα με κάποια διατύπωση, γιατί σήμερα εκεί σημειώνονται κάποια προβλήματα. Τώρα, έχω και ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο, σχετικά με μία παράγραφο όπου ο εισηγητής λέει για την ορατότητα και την ε, υλοποίηση ε, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Εδώ θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Τι ακριβώς ε, εννοούμε. Σταματώ εδώ και βεβαίως θα συνεχίσω να συνεργάζομαι εντατικά με τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ, σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Μαούρο και λυπάμαι που δεν αναφέρθηκε καθόλου ε, στους ασύριους χριστιανούς. Εν πάση περιπτώσει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο πέραν των ονομάτων θα έπρεπε να υπάρξει μια αναφορά στους ασύριους ε, χριστιανούς του Ιράκ. Ίσως θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε και σε άλλες θρησκευτικές μειονότητες όπως οι Γεζιντοί Νομίζω ότι οι χριστιανοί γενικότερα φύγονται ιδιαίτερα από τη σύγκρουση. Το 30% έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ή έχουν δολοφονηθεί. Μιλάμε για μια εθνοκάθαρση σε κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί. Λυπάμαι που αυτό δεν διευκρινίζεται ή δεν υπογραμμίζεται τόσο πολύ. Από ένα εκατομμύριο χριστιανούς στο Τικρίτ κάποτε τώρα είναι μόνο 300 ή 400 χιλιάδες. Όλοι υποφέρουν βέβαια στη χώρα αυτή, αλλά νομίζω ότι δυσανάλογα υποφέρουν οι ε, χριστιανοί. Να αναφερθώ επίσης στο δημοψήφισμα που έγινε στο Κυρκούκ, μια πόλη η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη λόγω των φυσικών πόρων που έχει. Νομίζω επίσης ότι στις προσθήκες ε, της δήλωσης της 6ης Οκτωβρίου δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διευκρινήσεις από τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν αυτοί οι οποίοι είναι υποπεριορισμό. Αν ο Αλμαλίκη θελήσει να τους, ε, ε, να στείλει στο Ιράκ, όλοι αυτοί θα εκτελεστούν νομίζω χωρίς ιδιαίτερες δικαστικές διαδικασίες. Πέραν αυτού υποστηρίζω την έκθεση. Κυρία Γκόμες, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ήμουνα η τελευταία εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα του Ιράκ Νομίζω ότι είμαι το άτομο που έχει ταξιδέψει πιο πολύ στο Ιράκ το τελευταίο καιρό. Ήμουνα εκεί πριν από δύο εβδομάδες, στο Ερμπίλ. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Μάουρο, τον Μάριο Μάουρο για την πολύ καλή του έκθεση. Ελπίζω θα μπορέσει να υπάρξει μια κοινή συμφωνία για ένα ψήφισμα για τη συμφωνία αυτή Πρέπει να σκεφτούμε στρατηγικά για το Ιράκ. Αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ. Και αυτή ήταν και η στάση του Κοινοβουλίου το 2008. Να σκεφτούμε τα συμφέροντά μας, τις αξίες μας. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει μονάχα σταθεροποίηση με τη μορφή που γίνεται στη Βόρεια Αφρική. Θέλουμε δημοκρατία, θέλουμε ένα ενωμένο, ομοσπονδιακό, δημοκρατικό Ιράκ και ο ρόλος μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τον εκτιμούν πάρα πολύ οι Ιράκινοι Κοιτάξτε ποια ήταν η ελεπίδραση του Ιράκ μαζί μας. Έχουμε την αντιπροσωπεία με το Ιράκ και τόσες φορές έχει έρθει ο αντιπρόεδρος και μέλη της αντιπροσωπείας αυτής από το Ιράκ εδώ και έχουν πει ότι θέλουν πράγματι να έχουν επαφές μαζί μας. Εμείς έχουμε κρατήσει μια επιφυλακτική στάση πολλές φορές γιατί κάποιες φορές δεν ήταν πολύ εύκολο να ταξιδεύσουμε στο Ιράκ λόγω της κατάστασης ασφαλείας. Όπω το αναγνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν με το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς για αυτά τα συμφέροντα. Το Ιράκ μπορεί να βοηθήσει να γίνει βιώσιμο το σχέδιο Ναμπούκο και, και δεν πρέπει να φοβηθούμε για κάτι τέτοιο. Επίσης υπάρχουν τεράστιες επιχειρηματικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν άλλοι στο Ιράκ αυτή το, η Τουρκία, η Κορέα, η Ινδία, η Ιαπωνία και είναι σημαντικό να υπάρξει διαφοροποίηση στην οικονομία του Ιράκ και εκεί τίθενται θέματα υδατίνων πόρων για τη γεωργία και χαίρομαι που στην περίπτωση της Τουρκίας είπαμε και κάποια για τη ροή του Τίγρη και του Εφράτη και τις συνέπειες για τη γεωργία και την ασφάλεια των περιοχών αυτών. Συμφωνώ λοιπόν με αυτούς που είπανε ότι η δημοκρατία μα ενδιαφέρει και αυτό σημαίνει πρέπει να έχουμε επαφή σε όλα τα επίπεδα μεταξύ κοινωνία των πολιτών, μεταξύ κοινοβουλίων κτλ. Πριν από δύο εβδομάδε ήμουν εκεί με την πρόσκληση του πρώην Υπουργού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράκ που έκανε μια <clears throat> συγκάλυψε μια συνδιάσκεψη γυναικών από τους ε, ΣΥΑ, τους Σουνίτες και τους Κούρδους. Και αυτό χρηματοδοτήθηκε ουσιαστικά από την Ιταλική κυβέρνηση. Και υπήρχαν και παρουσίες διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων. Όλα αυτά τα προβλήματα με τις γυναίκες, όπως είπε η Ελένη Κοπά, έχουν αντιμετωπιστεί σε αυτή τη συνδιάσκεψη. Μια τέτοια μορφή αλληλεπίδραση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να είμαστε σε επαφή με την πλειοψηφία του πληθυσμού στο Ιράκ, που είναι μια σαφή πλειοψηφία στο Ιράκ, γιατί τόσοι άντρε έχουν σκοτωθεί στην καταστολή του Σαντάμ και του πολέμου. Αν εστιάσουμε λοιπόν στα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράκ, θα προσφέρουμε μια μεγάλη υπηρεσία στο να εξασφαλίσουμε το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στο Ιράκ. Για τις μειονότητες, όχι μόνο τους χριστιανούς, αλλά και άλλες μειονότητες, πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν θύματα και στόχος τρομοκρατίας και ιδίω υπήρξε στόχος η χριστιανική μειονότητα. Δεν θα τους εξυπηρετήσουμε όμως ιδιαίτερα με το να έχουμε μια δυσανάλογη προσοχή για τους χριστιανούς, γιατί όλοι ήταν θύματα τρομοκρατίας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα σωστή, σωστό πλαίσιο για όλες τις μειονότητες και τα δικαιώματά τους. Το θέμα των φυλακών είναι πολύ σοβαρό. Και ιδίως οι φυλακές του Υπουργείου Εσωτερικών. Και φυσικά και η τύχη των κρατουμένων που είχαν συλληφθεί από τους Αμερικάνους και είχαν κάποια στιγμή φτάσει 26.000 και ήταν κρατούμενοι χωρίς κανένα νομικό πλαίσιο. Ίσως εκεί η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. <clears throat> Επίσης και το θέμα των ε, προσφύγων είναι πάρα πολύ σημαντικό και να αντιμετωπίσουν και το θέμα των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά, το οποίο είναι πολύ πιο οξύ από το πρόβλημα των προσφύγων. Εν κατακλείδη, χρειάζεται να ξεπεράσουμε τα προσκόμματα τα οποία υπάρχουν για να πάμε στο Ιράκ και συμφωνώ με αυτό που είπε και ο κύριο Κάτσιν ότι πρέπει να πάμε στο Ερμπίλ. Εγώ ήμουν εκεί πέρα πριν από δύο εβδομάδε. Κυκλοφορούσαμε το ταξί, πήγα στην ανοιχτή αγορά στο Σουκ και δεν με πήραξε κανένα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα αλληλεπίδραση με του Ιρακινού. Είναι παράλογο να μην μπορεί να πάει η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Έχουμε προξενία η Γαλλία, η Γερμανία, η το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ε, προξενία και έχουμε κατευθείαν πτήσεις από τη Γερμανία και την Αυστρία στο Ερμπίλ και μέσα στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αντιπροσωπεία μας στη Βαγδάτη θα πρέπει να έχει το δικό της κτίριο γιατί αυτό δεν έχει γίνει ακόμα και θα πρέπει να πιέσουμε για να υπάρξουν στενότερες σχέσεις μεταξύ της δικής μας αντιπροσωπείας και του Ιρακινού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάουρο λοιπόν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους που μου επιτρέπουν να εξηγήσω λίγο τη λογική η οποία βρίσκεται πίσω από αυτό το οποίο σας είπα. Σχετικά με ό,τι δεν προανέφερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που δεν είπα δεν είναι σημαντικά. Νομίζω ότι όλα μπορεί να είναι χρήσιμα ανάλογα με το επίπεδο φιλοδοξίας το οποίο έχουμε. Εμείς δεν κρύβουμε ότι θέλουμε να κάνουμε μια πλήρη ανάλυση της κατάστασης και να κάνουμε ξεκάθαρες προτάσεις. Όπως είπα το Ιράκ αυτή τη στιγμή ζει μια δύσκολη περίοδο και ακριβώς στα πλαίσια των σχέσεων που έχουμε με το Ιράκ εμείς νομίζω ότι θα πρέπει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπογραμμίσουμε το ποιες είναι οι συνθήκες πλέον εκδημοκρατισμού της ζωής της χώρας. Η συμφωνία αυτή δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε μια αυστηρά οικονομική αντίληψη, αλλά να έχει και πολιτικό περιεχόμενο. Συνεπώς λοιπόν, Η κυρία Κοπά πολύ σωστά είπε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να σημειώσουμε τις διακρίσεις τις οποίες υφίστανται όλες οι μειονότητες και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί της. Οι συνθήκες σεβασμού των δικαιωμάτων πρέπει να αφορούν τους πάντες και όλες τις μειονότητες και όλους τους πολίτες εν πάση περιπτώσει. Γιατί εγώ το κρύβω αν θέλετε λίγο αυτό ή επιμένω λίγο σε αυτά που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί. Είναι σαφές ότι έχει ξεκινήσει να προωθείται μία αντίληψη η οποία μετά από αυτά τα οποία έγιναν και στην Αλεξάνδρεια και μετά από τους χίλιους νεκρούς οι οποίοι έχουν σωρευτεί από πλευράς χριστιανών στο Ιράκ τον τελευταίο καιρό κάποιοι τρομοκράτες, κάποιες τρομοκρατικές ομάδες έχουν στην ουσία θέση σε ομοιρία τους χριστιανούς λέγοντας ότι επειδή είναι χριστιανοί είναι φιλοδυτικοί και φιλοαμερικανοί. Οι Ιρακινοί χριστιανοί όμως ανήκουν σε πολλές ομολογίες θρησκευτικέ, εκφράζουν έναν τεράστιο πλούτο και μια πολυπίκυλη πραγματικότητα προσεύχονται στην αραμαϊκή, στα συριακά, στα αραβικά, λατρεύουν τη χώρα τους και νομίζω ότι πρέπει να ονοματίσουμε το τέρας. Δεν πρέπει να δημιουργούμε προσπάθειες απομόνωσης και να τις τεκμηριώνουμε μέσα στην Ιρακινή κοινωνία. Θυμίζω ότι όταν έγινε η πρώτη απόπειρα εις βάρος της Κοπτικής Εκκλησίας στην Αιγύπτο, το Κοινοβούλιο παρενέβη αμέσως λέγοντας ότι ήταν μια επίθεση τρομοκρατική η οποία εμπνέεται από φονταμενταλιστές. Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση μας διέψευσε λέγοντας ότι ήταν θέμα οργανωμένου εγκλήματος και επίσης υπήρχαν και προβλήματα παράνομων σεξουαλικών σχέσεων κτλ. Αυτά ήταν φυσικά εντελώς εκτός θέματος. Βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να αποκρύψουμε την πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι οι χριστιανοί διαδηλώνουν σήμερα μαζί με τους αδελφούς μουσουλμάνους στην πλατεία του Καΐρου. Και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα ειδικότερο στην Ιρακινή πραγματικότητα, το ότι Ιδιαίτερα στις περιοχές του Κυρκού και της Μοσούλης ε, υποχρεώθηκαν να φύγουν, να πάνε στη Συρία, στην Ιορδανία. Υπάρχουν Ιρακινοί πρόσφυγες που θέλουν να παλινοστήσουν, θέλουν να επανενταχθούν στην κοινωνία τους και υπάρχει και ένα άλλο επιπλέον χαρακτηριστικό. Ο πρόεδρος Τζελάλ Ταλαμπάνι έκανε μία πρόταση έτσι ώστε να εντοπιστεί μία περιοχή η οποία να μετατραπεί ε, στην ε, πεδιάδα της Νινόβης σε ένα χριστιανικό έδαφος. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ιδιαίτερα σωστό, αλλά παρόλα αυτά το να μιλάμε για χριστιανούς δεν είναι μια προσπάθεια να τονίσω τη δική μου ταυτότητα. Να πω όμως ότι δεν μπορούμε εμείς να αγνοήσουμε την πραγματικότητα και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε τη συμβίωση όλων των κοινοτήτων, διότι είτε είναι χριστιανοί είτε δεν είναι, είναι κυρίως Ιρακινοί. Το δεύτερο ερώτημα που έθεσε η κυρία Κοπά έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κρίνουμε το πώς ε, λειτουργούν ορισμένες υπηρεσίες της νέας κυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί αυτά είναι ενδεικτικά της δημοκρατίας και της ποιότητας της δημοκρατίας. Πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο λοιπόν στο θέμα αυτών των υπηρεσιών και σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Κατσίν, ο οποίος παρατήρησε τη δυσκολία που υπάρχει να ολοκληρωθεί η κυβέρνηση γιατί υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε επίπεδο Υπουργείου Εσωτερικών και σε επίπεδο Υπουργείου Άμυνας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, μάχες για την εξουσία πάνω στις οποίες είναι δύσκολο προς το παρόν να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Τώρα, να πω επίσης ότι θα πρέπει να ευνοήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να γνωρίσουμε πραγματικά το τι κάνουν και σκέφτονται οι γυναίκες του Ιράκ για τη χώρα τους. Τι κινείται από τις γυναίκες αυτές τις χώρες, σε αυτή τη χώρα και τι είναι αυτό που είναι εμπόδιο στο να πρωταγωνιστήσουν στην Ιρακινή κοινωνία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία τώρα για τις συστάσεις τις οποίες έκανε η κυρία Μπρέπολς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί της. Υπάρχει άλλο ένα θέμα επίσης το οποίο αφορά την έκθεση αυτή είναι το θέμα των μέσων ενημέρωσης. Πρέπει να ζητήσουμε τα μέσα ενημέρωσης να είναι ανεξάρτητα και να δώσουμε εγγυήσει και αυτά για την καλύτερη συμβίωση των διαφορετικών κοινοτήτων στην χώρα αυτή. Οι παρατηρήσεις του κύριου Τάνοκ θα ληφθούν υπόψη. Νομίζω και μέσα από τις δικές του τροπολογίες και τις δικές μου θα συμπληρώσουμε το πλαίσιο της παρουσίασής μου. Και στα πλαίσια των επικοι... της επικοινωνίας που θα έχω και με τους κοιόδης εισηγητές και τους άλλους συναδέλφους δεν έχω κανένα με κανένα δισταγμό για να συμπληρώσω ε, τα θέματα με τα οποία ασχολείται η έκθεσή μου. Να κάνω εδώ μία αναφορά σχετικά με αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκόμες. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε να δώσω ε, ε, στην Επιτροπή μας τη δυνατότητα να πάει στο Ιράκ. Εγώ με κάθε ειλικρίνεια νομίζω ότι δεν υπάρχουν αξεπέραστα εμπόδια για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι και το θέμα της ασφάλειας θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρό τρόπο. Οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνουν στο Ιράκ, πηγαίνουν αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν, προετοίμασαν μάλλον τη συμφωνία Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ανοίξουμε λοιπόν ε, τις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Όπως λοιπόν τακτικά οι διάφορες διακοινοβουλευτικές επιτροπές ε, πηγαίνουν σε χώρες όπως ε, το Κουρδιστάν σε εισαγωγικά, νομίζω ότι θα ήταν ένα μήνυμα εμπιστοσύνης εμείς να πάμε στη χώρα αυτή και να δείξουμε ότι πιστεύουμε στην αναγέννησή της. Θυμίζω ότι κάποιες, κάποια δημοσιογραφικά πρακτορία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργάνωσαν εδώ και μία εβδομάδα εκτός της πράσινης ζώνης της Βαγδάτης μία ομάδα εργασίας για τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Αν τα κατάφεραν αυτά οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι από τις χώρες μας, γιατί να μην μπορέσει να τα καταφέρει ένα σημαντικό όργανο όπως το δικό μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο ακούστηκαν Προηγουμένω για, για τα χρονοδιαγράμματα. Εγώ είπα 16 Φεβρουαρίου. Γιατί? Εγώ δεν έχω επίσημη ενημέρωση από πλευρά του Συμβουλίου ότι δήθεν έχει κάποιες δυσκολίες να καταλήξει στη συμφωνία. Συνεπώ, εκεί όπου θα υπάρξει, όταν υπάρξει μια τέτοια επίσημη ανακοίνωση από πλευρά του Συμβουλίου, τότε θα μετακινήσουμε την προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών, αλλά μόνο τότε. Ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η πρόταση ψηφίσματο του κυρίου Πρέδα για την Ισλανδία. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Όπως ξέρετε, το... μέσα σε αυτό το... στην πρόσφατη Ολομέλεια εγκρίναμε το ψήφισμα σε σχέση με την αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο εβδομάδες μετά την έκδοση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου, τη σύσταση του Συμβουλίου που ζήτησε το, την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων, τι έχει γίνει έκτοτε λοιπόν σε επίπεδο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε η μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή καταρχήν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους Ισλανδούς συναδέλφους μας και τον Νοέμβριο ξεκίνησε η διαδικασία του screening της χώρας αυτής. Μέχρι στιγμής έχει γίνει το screening, η επισκόπηση 15 κεφαλαίων και το Μάρτιο θα είναι δυνατόν να έχουμε την έκδοση της πρώτης εκθέσεως για τα αποτελέσματα, τα πορίσματα του screening, κάτι το οποίο θα επιτρέψει, <clears throat> και είχαμε συζητήσει με τον Επίτροπο Φίλε για το θέμα αυτό, αυτό θα μπορούσε ίσως καταρχήν να επιτρέψει μέσα ακόμα στην Ουγγρική Προεδρία να ξεκινήσουν τα πρώτα κεφάλαια διαπραγματεύσεων. Για τα κύρια τώρα σημεία της έκθεσής μου έχω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα για τα πολιτικά κριτήρια είδαμε ότι υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι στην ε, ανεξαρτοποίηση της ε, δικαστικής εξουσίας. Βλέπω ότι κάποιοι συνάδελφοι είναι ακόμα στη συζήτηση για το Ιράκ. Δεύτερον, για τα οικονομικά κριτήρια. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο εδώ. Εμείς εργαστήκαμε επί τη βάση της προηγούμενης έκθεσης και εδώ πρόκειται για την ε, διαμάχη που υπάρχει μεταξύ της Ισλανδίας και των ε, και, της, ε, και των κάτω χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου για την υπόθεση ΑΣΕΙΒ. Αλλά αυτή η διαφορά τώρα νομίζω ότι έχει πάρει την οδό της επίλυσης. Είναι πολύ καλά αυτά τα νέα. Για τα οικονομικά κριτήρια επίσης, κάποιες ελλείψεις σε θεσμικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα έχουν ήδη ξεπεραστεί υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι για την εδραίωση ενός πλαισίου εποπτείας και ρυθμίσεως στον χρηματοοικονομικό τομέα. Και επίσης για τα οικονομικά θέματα και πάλι <clears throat> ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι βγήκε από την ύφεση η Ισλανδική οικονομία. Αυτό είναι πολύ θετικό. Έχει βγει τελείως από την ύφεση. Τρίτο κεφάλαιο το οποίο θέλω να θίξω, εν συντομία, το θέμα της κοινή γνώμης. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια ευρεία πλειοψηφία, 65% των Ισλανδών, υπέρ της ένταξης της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, το Ισλανδικό Κοινοβούλιο στην Ρέικ Γιαβίκ έχει το στόχο να ξεκινήσει μια ευρεία εκστρατεία πληροφόρησης για τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ώστε οι Ισλανδοί πολίτες να μπορούν στο τέλος του, της διαδικασίας να επιλέξουν εάν θέλουν πράγματι να λάβει χώρα αυτή η είσοδος της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον και αδημονία τις συνεισφορές όλων των συναδέλφων για τη βελτίωση αυτής της έκθεσης 16 Φεβρουαρίου <clears throat> είναι καταληκτική προθεσμία για την ε, κατάθεση τροπολογιών και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ λέει και ο κύριος Δεν βλέπω να... Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Πεντά μας είπε ότι η προθεσμία των τροπολογιών είναι 16 Φεβρουαρίου και για την Μακεδονία, η πρώην Μακεδονία ήταν 15 Φεβρουαρίου. 16 λοιπόν για την Ισλανδία, 15 για την Πουδουγούμου. Έχουμε τώρα μια αντιπροσωπεία από την ακτή του Ελεφαντοστού, τον κύριο Γουαταρά, τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας αυτής. Είναι μια ακρόαση που κάνουμε μαζί με την Επιτροπή Ανάπτυξης και μαζί με την ισομερή συνέλευση ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Τζετζέ Μαντί είναι μαζί μας, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος της ε, Ακτής του Ελεφαντοστού. Δεν είναι παρούσα ακόμα όλη η αντιπροσωπεία. Λίγη υπομονή παρακαλώ.

Ο κ. Μαχτή, ο Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος Κωτιβουάρ είναι μεταξύ μας και σας δίνω μέσα στον λόγο. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αγαπητά λοιπόν μέλη, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα εξ ονόματος του Προέδρου Αλασάν Ντραμάν Ουαταρά, της κυβέρνησής του και της Δημοκρατίας της Κοντιβουάρ να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει από τότε που ξέσπασε η κρίση στη χώρα μου το 2002 έχετε υποστηρίξει τη χώρα μου σαν Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς ιδιαίτερα στον τομέα της οργάνωσης ε, της κατάστασης για την έξοδο από την κρίση και της χρηματοδότησης που ήταν απαραίτητη. Ήσασταν παρόντες επίσης και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της εκλογικής διαδικασίας μέσω των παρατηρητών σας, οι οποίοι είδαν το πώς πήγαν τα πράγματα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας με τις χώρες ΑΚΕ που ήδη από την 3η Δεκεμβρίου αντέδρασε σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μου. Είναι σαφές ότι η κρίση την οποία ζει η χώρα μου εδώ και 10 χρόνια σχεδόν είναι καταρχάς μια κρίση εμπιστοσύνης Ήδη από το 2005 με τη δεύτερη συνάντηση της Πρετόρια και μετά από αίτημα του Ουαταρά εκείνη την εποχή είχε πει ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε το θέμα της εξόδου από την κρίση με δημοκρατικό τρόπο ελεγχόμενο από τα Ηνωμένα Έθνη. Εκείνη την εποχή ο προεδρεύων της χώρας μου, ο Λορόν Μπαγκμπό, πρότεινε την λύση και πρόκρινε τη λύση της διαιτησίας από πλευρά της διεθνούς κοινότητας μέσω μιας επιτροπής πιστοποίησης των αποτελεσμάτων. Και έτσι η ευρωπαϊκή ή η διεθνής κοινότητα μάλλον προσπάθησε να μας βοηθήσει και όταν ξεκίνησε η αντιμετώπιση των προβλημάτων δυστυχώς υπήρξαν πολλά προβλήματα τα οποία προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε μέσω της βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών και της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών και φτάσαμε στη δεύτερη φάση στον κατάρτιση των λεγόμενων λευκών καταλόγων εκλογικών καταλόγων ε, θέλησαμε να υπάρξει επιστοποίηση από πλευράς της διεθνούς κοινότητας μέσω του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κάτι το οποίο κατέστησε έγκριτες τις λύσεις αυτές, οι οποίες έγιναν δεκτές από τους 14 υποψηφίους πρόεδρους. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν εξελίχθηκε και ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας που οδήγησε στον δεύτερο γύρο τον Μπαγμπό και τον Ουαταρά. Υπήρξε ένα πρόβλημα σε σχέση με την ανάγνωση των αποτελεσμάτων στο δεύτερο γύρο. Ήδη από τον πρώτο γύρο αυτό το οποίο ζητήθηκε από την Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή ήταν η μετάδοση όλων των εκλογικών εγγράφων τρεις ημέρες μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας και όχι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Και έτσι μετά από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων τα έγγραφα ταξινομήθηκαν σε επίπεδο ε, περιφερειών ή νομών και απεστάλησαν στην Κεντρική Επιτροπή στον διαμεσολαβητή της Αφρικανικής Ένωσης, τον κύριο Καμπαόρε, στον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών και στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε 72 ώρες. Σχετικά με την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την ανακοίνωση μέσα σε 72 ώρες. Κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή έγινε την τέταρτη μέρα στις 2 η ώρα το πρωί και αυτό δεν προκάλεσε καμία ιδιαίτερη δυσκολία σε αυτήν την διαιτησία από πλευρά του διαμεσολαβητή και πιστοποιητή. Αυτό έγινε μετά από την έκδοση της απόφασης του Συνταγματικού Συμβουλίου. Και έτσι βρεθήκαμε λοιπόν στον δεύτερο γύρο και κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου ξεκαθαρίστηκε ότι ο κυρίαρχος λαός της χώρας μου ψήφισε κατά πλειοψηφία κατά 54,10% υπέρ του Ουαταρά και ο Ουαταρά εξελέγει πλέον πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κοντιβουά. Εν τω μεταξύ, το σύνολο της διεθνούς κοινότητας παρακολούθησε το τι έγινε κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας της καταμέτρησης όπου οι εκπρόσωποι του Προέδρου Μπακμπο στα πλαίσια μιας πλήρους ατμόσφαιρας ανασφάλειας ήρθαν να πάρουν από τα χέρια του εκπροσώπου της Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής το έγγραφο το οποίο ανακοίνωνε τα προσωρινά αποτελέσματα και έτσι και ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής ο Ιουσούφ Μπακαγιόκο για λόγους ασφαλείας πήγε στο λεγόμενο Grand Hotel της, του Αμπιτζάν και ανακοίνωσε εκεί τα αποτελέσματα. Να θυμίσουμε επίσης και το τι προβλέπει το άρθρο 64 του εκλογικού κώδικα. Προβλέπεται όπου στην περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσμα που ανακοινώνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή αμφισβητηθεί από το Ανώτατο Συνταγματικό Συμβούλιο, τότε ακυρώνονται αυτές οι εκλογές που ήσαν εν αμφιβολία και η Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή έχει 45 ημέρες για την αναδιοργάνωση των εκλογών. Το Συνταγματικό Συμβούλιο σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα και την εξουσία να ακυρώσει ένα τμήμα των εκλογών και να ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα επί τη βάση μόνο ενός τμήματος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, Βλέπουμε ότι ήδη είχαμε να κάνουμε με τον πρόλογο ενός στρατιωτικού κινήματος το οποίο ήθελε ο Κμπακμπό να οργανώσει. Σε επίπεδο δημοκρατίας λοιπόν είναι σαφές ότι ο πρόεδρος που εξέλεξαν οι κάτοικοι της χώρας μου είναι ο Ντραμαν Ουαταρά και θέλω να ευχαριστήσω τη διεθνή κοινότητα, από την Αφροκανική Ένωση, από την Ένωση Οικονομικής Συνεργασίας Δυτικής Αφρικής και τα Ηνωμένα Έθνη, που μέσω των παρατηρητών τους, μέσω επίσης των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα του Ιδίου, μέσω των προσπαθειών που έκανε ο Καμπαορές σαν διαμεσολαβητής, αναγνώρισαν στο τέλος της διαδικασίας τον Ουαταρά σαν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από τότε λοιπόν που αυτό το δημοκρατικά, δημοκρατικό αποτέλεσμα είναι γνωστό, τι βλέπουμε. Βλέπουμε να διαφημίζεται η βία. Ο πρόεδρος Μπαγκμπο είπε ότι είχε πέσει θύμα στρατιωτικού πραξικοπήματος το 2002, δεν αποχωρεί σήμερα και χρησιμοποίησε στρατιωτικές δυνάμεις εις βάρος του δημοκρατικά εκλεγμένου Ουαταρά. Έτσι λοιπόν είμαστε μάρτυρες ενεργειών βίων, 370 νεκροί. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ περισσότεροι. Αυτοί έχουν αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Και σε καθημερινή βάση έχουμε νέα αθώα θύματα της βαρβαρότητας και της επιθυμίας του Μπακμπό να γατζωθεί στην εξουσία μέσω της βίας. Την προηγούμενη εβδομάδα φαντάζεστε ότι στην πόλη του Αμπιτζάν μόνο δύο δήμοι αυτή τη στιγμή υπόκεινται ε, σε απαγόρευση κυκλοφορίας εδώ και δύο μήνες. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια προσπάθεια καταστολής ε, των κινημάτων των πολιτών. Καταστράφηκαν και δύο αστυνομικοί σταθμοί επειδή ε, δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του Κμπάγκμπο. Έκανε προσπάθειες η διεθνής κοινότητα, υπήρξε ένα πάνελ του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας το οποίο κατέληξε χθε σε συμπεράσματα και είμαστε πεπισμένοι ότι ο κύριος Μπακμπό δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διάθεση σεβασμού της δημοκρατίας και δεν σκοπεύει να αποσυρθεί μετά από την εκλογική του ήττα. Κάθε μέρα συσσωρεύονται και περισσότεροι νεκροί στη χώρα μου και γι' αυτό θέλω να ζητήσω από τη διεθνή κοινότητα να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα ανθρωπιστικής παρέμβασης, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν όλο και περισσότεροι άμαχοι, αθώοι, οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στις διάφορες γειτονιές του Αμπιτζάν και στο εσωτερικό της χώρας μας. Ο πρόεδρος Παταρά και το κόμμα μας, το Δημοκρατικό Κόμμα και το Συνασπισμός για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία που του οποίου ηγήθη θέλουν μια λύση μετά από διαπραγματεύσεις. Αλλά θέλουμε να δούμε την, πρέπει να δείτε την πραγματικότητα όπως είναι. Η διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει για όλα τα θέματα εκτός από ένα. Ζητάμε ανεφόρον όπως προέκυψε από την κάλπη να αναγνωρίσει ο πρόεδρος Μπαγμπό την νίκη του κυρίου Βαταρά και να μπορέσει να εγκαθιδρυθεί ο κύριος Βαταρά και να ασκήσει το δημοκρατικό του αξίωμα. Όλα τα άλλα μπορούν να συζητηθούν και να τύχουν διαπραγμάτευση. Και εξάλλου, να σα υπενθυμίσω στην τελευταία συνεδρία του Συμβουλίου Συνεργασίας της Δυτική Αφρικής στο Ουαντουγκουντού, ο πρόεδρος ε, και ο κ. Βαταρά ήταν παρόντες και είπαν ότι όποιο κερδίσει τι εκλογέ προ το συμφέρον τη ε, του ελεφαντοστού προς το συμφέρον της συμφιλίωσης θα σχηματίσουν μια κυβέρνηση η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις συνιστώσεις και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ώστε να μπορέσει να οικοδομηθεί η ειρήνη στη χώρα μου, να ενισχυθεί η εσωτερική μας συνοχή και να προχωρήσουμε προς την ανάπτυξη της χώρας μας. Αλλά είναι γεγονός ότι η Κοντιβουάρ δεν μπορεί να χωριστεί στα δύο, ότι η χώρα αυτή δεν μπορεί να έχει δύο προέδρους και ότι ο λαός της ε, ακτής του Ελεφαντοστού έχει ένα πρόεδρο, τον Άντρασαν Ουαταρά. Πρέπει να αναγνωριστεί το αποτέλεσμα της, των εκλογών και πιστεύουμε ότι η διεθνή κοινότητα η οποία συμμετείχε από την αρχή ως το τέλος σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ να γίνουν τα απαραίτητα, οι απαραίτητε ενέργειε για να αναγνωριστεί η νίκη του Ουαταρά και να αναλάβει την εξουσία. Κυρίε και κύριοι, ως εκπρόσωποι της ε, ακτής του ελεφαντοστού βασιζόμαστε στην διεθνή κοινότητα, γιατί είμαστε και εμείς ένα μέλος της διεθνούς κοινότητας κρατών και εθνών. Στο βαθμό που η θέση του Πρόεδρου Μπακμπό είναι να διατηρήσει την εξουσία πάση και με τη βία, η διεθνή κοινότητα δεν θέλει να δει να λαμβάνει χώρα μια νέα Ρουάντα και επομένως για να αποτρέψει κάτι τέτοιο θα πρέπει να παρέμβει ώστε να γίνει σεβαστή η δημοκρατία. Κάνουμε μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένα από τα σημεία αναφοράς για όλους τους δημοκράτες στον κόσμο να πράξει τα απαραίτητα ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το οποίο έγινε στην ε, ακτή του Αλεφαντοστού και να μην υπάρξουν μιμητές της. Γιατί εάν όλοι οι τιμένοι πρόεδροι στην Αφρική θα μείνουν στην εξουσία με την υποστήριξη του στρατού, τότε μπορούμε να ξεχάσουμε τη δημοκρατία στην Αφρική. Όλοι μας θα πρέπει να αγωνιστούμε για να υπάρξει πλήρης σεβασμός της δημοκρατίας και για να υπάρξει σεβασμός της δημοκρατίας θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα πάρει την προεδρική εξουσία κ. Γουαταρά. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσει η διεθνή κοινότητα να τον αναγνωρίζει ως μόνο νόμιμο πρόεδρο και να επιτρέψει στην Κορτιβουά να είναι ένα δημοκρατικό έθνος μεταξύ όλων των άλλων και σας ευχαριστώ για την προσοχή που δώσατε στα λεγόμενά του και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να έλθουμε ενώπιόν μας εξ ονόματος του Πρόεδρου Αλασάν Ουαταρά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα, καλώς ήλθατε και ευχαριστώ όλη την αντιπροσωπεία σας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Στασνή, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μικτή Επιτροπή ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε... Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα αγγλικά, πιο εύκολο θα είναι για μένα. Ο συμπρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ο Λουί Μισελ, δεν μπόρεσε δυστυχώς να παρευρεθεί σε αυτή τη σημαντική συνάντηση θα απευθυνθώ στην αντιπροσωπεία του Προέδρου της Ακτής του Αλεφαντοστού ως αντιπρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, η οποία παρακολούθησε εκ του σύνεγγης της εξελίξεις στην ακτή του Αλεφαντοστού ε, κατά τη διάρκεια και μετά τις πολιτικές εκλογές στα τέλη του περασμένου έτους. Επιτρέψτε μου επίσης να υπογραμμίσω ότι η συνέλευση ήταν ε, από τα πρώτα κοινοβούλια που αντέδρασαν στην ε, κατάσταση μετά τις εκλογές στη χώρα στις 4 Δεκεμβρίου στην 24η ε, συνεδρίασή της στην Κινσάσα ενέκρινε δήλωση σχετικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στην ακτή του Ελεφαντοστού. Στη δήλωση αυτή ε, δήλωσε την, ε, τον αποτροπιασμό της για τις ταραχές στη χώρα που οδήγησε σε θύματα ε, όταν ανακοινώθηκαν προσωρινά αποτελέσματα. Καταδίκασε επίσης την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου να ακυρώσει τα προσωρινά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν από ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή της ακτής του Ελεφαντοστού. Όπως υπογραμμίζει η δήλωση, η μεικτή συνέλευση αρνείται να δεχτεί τα αποτελέσματα που έδωσε το Συνταγματικό Συμβούλιο γιατί θεωρεί ότι ε, δεν εκφράζουν τη βούληση του λαού της χώρας. Θα ήθελα να τονίσω ότι για την ε, συνέλευσή μας ως Δημοκρατικό Κοινοβούλιο το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ο σεβασμός της βούλησης του λαού της χώρας. Ε, από το 2005 ε, προσπαθεί ο λαός να δηλώσει την βούλησή του και την προτίμησή του από ό,τι φαίνεται στον πρόεδρο Ουατάρα. Κατανοούμε τον κίνδυνο από τη σημερινή κατάσταση στην πολιτική και κοινωνική ισορροπία που με δυσκολία επετεύχθη στην ακτή του ελεφαντοστού και τη σταθερότητα σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η ομάδα που συστάθηκε τέλος Ιανουαρίου από το Συμβούλιο Ασφάλειας και Ειρήνης ε, για να αντιμετωπίσει την κρίση στη χώρα ε, επέτυχε να βρει, εξεύρει την καλύτερη λύση στο πρόβλημα της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πέντα, ο οποίος είναι επικεφαλής, ήταν επικεφαλής της ε, ομάδας παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εκλογές. Θέλω να επιμείνω στο θέμα αυτό των εκλογών. Είχαμε συζητήσει ήδη πριν από δύο εβδομάδες για το θέμα αυτό, όταν είχε παρουσιαστεί επίσημα η έκθεση για τις εκλογές. <clears throat> Θέλω να υπογραμμίσω τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα. Το πρώτο το ανέφερε ο κύριος ε, Μάντι, ο υπουργός κύριος Μάντι, είναι κατάσταση που είναι μια κατάσταση ουσιαστικά εμφυλίου πολέμου που γνωρίζει τώρα η ακτή του Κότ Ντιβουάρ. Εκατοντάδες νεκρών. Πολλοί κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση, κατάσταση όπου κινδυνεύει η ζωή του. Πολλοί απειλούνται αυτή τη στιγμή Υπάρχει τεράστια λοιπόν ανασφάλεια η οποία σοβεί στην χώρα αυτή και δεν απέχουμε πολύ από ένα πραγματικό εμφύλιο πόλεμο εκεί. Οι συνθήκες λοιπόν απέχουν πολύ από τις φυσιολογικές συνθήκες. Δεύτερον, θέλω να τονίσω ότι υπάρχει απόλυτα άκαμπτη στάση του Προέδρου Μπαγκμπό. Ήδη από το δεύτερο γύρο αρνήθηκε να μετακινηθεί ούτε κατά ένα χιλιοστό. Εξακολουθεί να κρατάει την θέση που είχε και προηγουμένως και επομένως αυτοί οι οποίοι περιμένουν ακόμα να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και από τις διαπραγματεύσεις αυτές να μπορεί να υπάρξει κάποια κίνηση, νομίζω ότι εισφάλουν. Εγώ έχω μεγάλο σκεπτικισμό σε σχέση με την δυνατότητα αυτές οι διαπραγματεύσεις να μπορέσουν να καθορίσουν να οδηγήσουν σε μια πιο ορθολογική αντιμετώπιση του κυρίου Μπακμπό. Και εξάλλου η αποτυχία των διαπραγματεύσεων και της διαμεσολάβησης θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο του κυρίου Μπακβό. Θα πιστεύει ο κόσμος ότι εφόσον αντέχει ακόμα, θα αντέξει για πάντα. Άμα αποτύχουν λοιπόν οι διαπραγματεύσεις, αυτό θα είναι προς όφελος του κ. Μπαγμπό. Και ένα τρίτο σημείο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω έχει να κάνει με τη θέση των αφρικανικών χωρών. Αν στην Ευρώπη υπήρξε τέλεια αλληλεγγύη και ταχεία αντίδραση σε σχέση με την κατάσταση στην ακτή Ελφαντοστού, Μπορεί στην αρχή να υπήρξε απόλυτη συνένεση, στη συνέχεια αυτή η συνένεση δεν υπάρχει πλέον. Ήμουνα στην ε, Αμπούτζα με την ε, Επιτροπή Συνεργασίας για τη Δυτική Αφρική και είπε ότι αυτή η σύγκρουση ε, φέρνει αντιμέτωπες χώρες της Δυτικής Αφρικής με την Νότια Αφρική, η οποία Νότια Αφρική προσπαθεί να επιβάλλει στην περιοχή αυτή της Δυτικής Αφρικής την επιρροή της. Προσπαθεί η Νότια Αφρική να περάσει τις δικές της γραμμές σε σχέση με τα θέματα αυτά. Πρέπει να δούμε λοιπόν ότι υπάρχουν μεγάλες εντάσεις μέσα στην Αφρικανική Ήπειρο τη στιγμή αυτή που ένα πάνελ αρχηγών κυβερνήσεων της Αφρικής προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι θα γίνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Το μόνο ερώτημα που έχω να θέσω στον κύριο Μαντή είναι το αν θεωρεί ότι μία στρατιωτική επέμβαση θα γίνει αναπόφευκτη αν και αυτή η προσπάθεια διαμεσολάβησης αποτύχει. Ή κατά πόσον θεωρείται ότι θα πρέπει συνεχιστούν οι προσπάθειες διαμεσολάβησης όλο το 2011. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Κάποιο άλλο θέλει να λάβει το λόγο. Κύριε Γενική Γραμματέα. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για μια αντικειμενική παρουσίαση την οποία έκανε. Νομίζω ότι με ρεαλιστικό τρόπο παρουσίασε την κατάσταση που μας απασχολεί. Δυστυχώς συμμερίζομαι την απεσιοδοξία του για τα αποτελέσματα της αποστολής υψηλού επίπεδου την οποία έχουν αναλάβει οι εκπρόσωποι αυτών των χωρών στην Κοντιβουάρ. Δεν περιμένουμε πολλά θα πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι σήμερα ήδη στο Αμπιτζάν το στρατόπεδο του Μπακμπό οργανώνει διαδηλώσεις για να πιέσει και να αρνηθεί την συμμετοχή στο πάνελ κάποιων μελών της ε, οργάνωσης για την Αφροκανική Ενότητα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Αν δεν υπήρχαν θάνατοι, αν δεν υπήρχαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Κάθε μέρα που περνάει δυστυχώς όμως μια τέτοια προοπτική δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή. Αυτό που είναι σαφές επίσης είναι ότι ο πρόεδρος Μπάκμπο θέλει να διατηρηθεί στην εξουσία μέσω της βίας. Γνωρίζετε και δεν χρειάζεται ίσως να το θυμίσω ότι ο πρόεδρος Μπάκμπο, ο οποίος είχε πάρει μέρος στο ε, πραξικόπημα του 2002 και θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να το κάνει αυτό και εις βάρος εκ νέου του Αταρά. Βρίσκεται σε μια λογική η οποία λέει ότι ο Αταρά απέτυχε το 2002 μεν, ο ίδιος επειδή έχασε τις εκλογές κάνει το δικό του πραξικόπημα βασιζόμενο στον τακτικό στρατό και στα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του ληστεύοντας ε, τη Θηγατρική Τράπεζα της Ένωσης Δυτικής Αφρικής, απαιτώντας ε, πληρωμή λίτρων από κάποιες άλλες χώρες ε, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσει του. Λοιπόν, εφόσον θέλουμε να υπάρξει μια λύση, αναβάλλοντας για κάποια περίοδο μια στρατιωτική επέμβαση η οποία φαίνεται να είναι αυτοεπιβαλόμενη αν πολλής, θα πρέπει ο κύριος Μπακμπό θα πρέπει να κατανοήσει ποιος είναι ο ρόλος του και γι' αυτό σε μια πρώτη φάση όπως είπα σας ευχαριστούμε και για την οικονομική σας βοήθεια αλλά όταν δεν θα έχει χρήματα ο Μπακμπό για να πληρώσει τους μισθοφόρους, τις πολιτοφυλακές, τους στρατιώτες οι οποίοι υφίστανται αυτή την άδικη αποστολή που πιστεύουν ότι το κάνουν για τη χώρα τους. Και υπάρχει και το θέμα της συμπεριφοράς, αν θέλετε, του στρατού, που βασίζεται ο Μπακμπό και ασκεί βία εις βάρος του πληθυσμού μέσω του στρατού. Ένα στρατός ο οποίος δεν είναι σαφώς υπέρ, αλλά τρία βασικά τμήματα, τα οποία όμως είναι ένοπλα, ισχυρά, ασκούν βίες ενέργειες εις βάρος του πληθυσμού. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο εξοπλίζονται καλύτερα, και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τα όργανα που είναι σε καλύτερη θέση από μένα για να γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται με το εμπάργο όπλων που είχε επιβληθεί στην Κοντιβουάρ γιατί συνεχίζει μέσω της Αγγόλα να εξοπλίζει τον Μπακμπό και στο εσωτερικό της Οργάνωσης Αφρικανικής Ενότητας ακούγονται και άλλες φωνές. Υπάρχουν πολλοί ε, οι οποίοι ζηλεύουν τον Μπακμπό και πιστεύουν ότι στο μέλλον θα μπορέσουν να ε, κάνουν και αυτοί τα ίδια που κάνει ο Μπακμπό όταν έρθει η σειρά τους εις βάρος της βούλησης ε, του πληθυσμού. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι δυστυχώς πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό η στρατιωτική παρέμβαση φαίνεται να είναι ε, προφανής πλέον ανάγκη. Νομίζω ότι προετοιμάζεται ο ίδιος ο πρόεδρος Πακμπό για μια τέτοια σύγκρουση γιατί πέρα από τον οπλισμό τον οποίο ε, προχωρεί να αγοράζει υπάρχει στράτευση πληθυσμού σε όλη τη χώρα όπου πολλοί άεροι γυναίοι προσλαμβάνονται σε εισαγωγικά για να πάνε στο στρατό, τους ε, εκπαιδεύουν για μία εβδομάδα μόνο και τους δίνουν καλάσνικοφ για να σκοτώσουν και να σκοτωθούν. Λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επαναλαμβάνω ότι στα πλαίσια αυτής της πραγματικότητας ε, το δικαίωμα ανθρωπιστικής παρέμβασης της διεθνούς κοινότητας είναι απαραίτητο να γίνει πραγματικότητα και αυτό για να τεθεί τέλος στο δράμα το οποίο ζει ο άμαχος πληθυσμός. Αυτός ο άμαχος πληθυσμός που πυροβολείται σε κάθε διαδήλωση με πραγματικές σφαίρες και δυστυχώς καθημερινά προστίθενται νεκροί σε αυτή την προσπάθεια. Αν μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό χωρίς στρατιωτική παρέμβαση γιατί όχι, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση με τον ελάχιστο δυνατό παράπλευρο απολειών. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπερμαντ από την Επιτροπή Ανάπτυξη για να κλείσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο είναι παράδοξο είναι ότι στη Γαλλία όταν είναι κανείς πρόεδρος μια μέρα παραμένει πάντα πρόεδρος. Τον αποκαλούν όλοι κύριε Πρόεδρε μέχρι το θάνατό του. Και κάποιοι το παίρνουν αυτό το θέμα πολύ στα σοβαρά, φοβάμαι. Νομίζω ότι ο Λοράν Παγμπό θα πρέπει να κατανοήσει ότι έχει σταθεί πρόεδρος και αυτό είναι μια μεγάλη τιμή. Αλλά αυτό ανήκει πια στην ιστορία. Έχει τελειώσει. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σωστά έπραξε να πάρει μέτρα <clears throat> χρηματοοικονομικών περιορισμών και περιορισμών για την ε, τι προξενικές θεωρίες. Πρέπει να εμποδίσει λοιπόν αυτές τις ολιστήσεις κύριε Μάντι και θα πρέπει να εμποδίσει τις προσπάθειες του κυρίου Μπακμπό και του του ο οποίος προσπαθεί να εκβιάσει αυτή τη στιγμή και θέτει την χώρα του σε κίνδυνο <clears throat> εμφυλίου πολέμου. <clears throat> Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να εξασφαλιστεί η ενότητα της χώρας αυτής και το να εξοπλίζεται δεν βοηθάει καθόλου. Αλλά ο κ. Παγκμπό εξακολουθεί να είναι παρόν χωρίς καμία νομιμοποίηση θεωρεί ακόμα τον εαυτό του πρόεδρο, ακόμα και όταν δεν τον αναγνωρίζει κανείς. Ούτε μια χώρα στον κόσμο δεν τον αναγνωρίζει. Μιλάμε για μια συνωμοσία, μιλάμε για γενική παράνοια η οποία ισχύει εκεί. Εμείς πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε τη δημοκρατική θέληση του λαού της ε, Κοντιβουάρ όπως έχει διαδηλωθεί από όλο τον κόσμο. Στην αρχή ήταν πολύ καλή η αντίδραση της, ε, Αφρικανική, της Ένωσης για την Αφρικανική Ενότητα, όπως επίσης και της Ένωσης των κρατών της Δυτικής Αφρικής. Σήμερα όμως φαίνεται ότι αυτή η στεναρή σχέση, στάση έχει αποδυναμωθεί. Αυτό κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν στρατηγικά συμφέροντα για την ενίσχυση της Αφρικανικής Ένωσης για να υποστηρίξει τα συμφέροντα και τη θέληση των λαών της Αφρικής για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η δημοκρατία στις χώρες αυτές. Και είναι κάτι το οποίο αποτελεί και στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχυθεί η Αφρικανική Ενότητα προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς θα πρέπει να σταματήσουμε να αναγνωρίζουμε τους δικτάτορες όπου μας βολεύει, όπως έγινε στην Τινησία, στην Αίγυπτο, και σε άλλες χώρες. Και φυσικά, και δεν μπορούμε να το πράξουμε αυτό στην ακτή του αλεφαντοστού. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει την πίεση σε χώρες όπως η Αγγόλα που παίζουν το παιχνίδι αυτό το, ε, το πολύ αρνητικό με το να δίνουν εξοπλισμό στον κύριο Μπάνγκμπο. Οι ενέργειες αυτές οι οποίες έχουν γίνει στις, ε, μετά από τις εκλογές ήταν Χωρί προηγούμενο, γιατί στην Κένια εξακολουθούν οι προσπάθειε να υπάρξει κάποια συμβιβαστική λύση, αλλά στη δική σα περίπτωση θα πρέπει να αναγνωριστεί η δημοκρατική θέληση. Και δυστυχώ, αυτή τη στιγμή υπαναχωρούν πάρα πολύ. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει τον ρόλο τη, θα πρέπει να δώσει δυνατότητα στην Αφρικανική Ένωση να παίξει τον πρώτο ρόλο και να ασκήσει τη διπλωματική πίεση η οποία είναι απαραίτητη αλλά εμείς θα πρέπει να είμαστε πάντα παρόντες σε αυτή τη διαδικασία και να μην μειωθεί καθόλου η ευρωπαϊκή πίεση. Αλλά δεν θέλουμε εμείς να είμαστε οι πρώτοι και οι πιο ορατοί και να δεχθούμε κατηγορίες για νεοαπικιακό τρόπο συμπεριφοράς. Ενώ οι αφρικανικές ενώσεις θα πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο. Χαίρομαι λοιπόν για την παρουσία σας και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα σας βοηθήσουν στον αγώνα σας στην Κωτιβουάρ. Ευχαριστώ, λέει και ο κύριος Μπόντης. Πριν κλείσουμε, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω. Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Ουαταρά και ο Πρωθυπουργό ο κύριος Σόου και οι αρχές της χώρας γύρω από τον πρόεδρο Ουαταρά εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες σε αυτό το, το περιορισμένο χώρο. Μήπως θα μπορούσατε να σκεφτείτε να πάτε στο Γιαμουσουκρό, στην πολιτική πρωτεύουσα, όπου θα βρείτε θα έλεγα μια ελευθερία πολιτικής δράσης την οποία σας στερούν στο Αμπιτζάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το να πάμε στο Γιαμουσουκρό είναι στόχος της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Ουαταρά. Είχε πει ότι αν εκλεγεί θα εγκαταστεθεί στο Ιαμουσούκρο. Και από εκεί θα προχωρήσει στην μεταφορά της διοικητικής πρωτεύουσα. Σήμερα όμως οι συνθήκες δεν προσφέρονται για κάτι τέτοιο. Γιατί κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες το να πάει στο Γιαμουσουκρό στην ουσία είναι σαν να επικυρώνει τον διαχωρισμό της χώρας, τη διαίρεση της χώρας. Αν αναγνωρίσουμε εμείς την δημοκρατική εκλογή του αλλά σαν Ουατάρα σαν Προέδρο το πρώτο καθήκον του είναι να διασφαλίσει την ένωση της χώρας έτσι ώστε η Κοντιβάρ να παραμείνει μία και αδιέρετη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το να πάει στο Γιαμουσουκρό θα είναι χειρότερο γιατί θα οδηγήσει στη διέρεση της χώρας για ολόκληρες δεκαετίες. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε να γίνουν ό,τι είναι δυνατόν και σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο έτσι ώστε ο Λορόν Μπακμπό να κατανοήσει. Όπως είπε ο εισηγητής σας, να κατανοήσει λοιπόν ότι ήταν πρόεδρος και μπορεί να παραμείνει πρόεδρος. Θα τον ονομάζουμε πάντα πρόεδρο, όπως ακόμα και όταν είσαι σε διοικητικά συμβούλια φοιτητικά. Μια φορά πρόεδρος, μένεις πρόεδρος για πάντα, αλλά δεν μπορεί η Κοντιβουάρ να παραμείνει κατά από τις σημερινές συνθήκες. Ιδιαίτερα επειδή και ο Ουαταρά πιστεύει στην πολιτική του Φελίξ Χουφουέτ Μπουανί, πιστεύουμε να υπάρξει ειρήνη έτσι ώστε όλοι οι κάτοικοι και του Βόρα και του Νότου και της Δύσης και της Ανατολής της Κοντιβουάρ να συνεργαστούν και να οικοδομήσουν μια Κοντιβουάρ με κάποιες δυνατότητες εξυπηρέτησης και των δικών συμφερόντων και των συμφέροντων της περιοχής για να μπορέσει να λειτουργήσει σαν κινητήρια δύναμη της περιοχής. Θυμίζει ότι από την αρχή όταν είχαμε πάει στο Μαρκουσί για τις πρώτες διαπραγματεύσεις τέθηκε στο κεφάλαιο 7 η κρίση της Κοντιβουάρ, δηλαδή μια κρίση η οποία θέτει εν κινδύνο την περιφέρεια, την ειρήνη στην περιφέρεια και την παγκόσμια ειρήνη. Αυτό λέει το 7ο κεφάλαιο της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, εμείς δεν επιδιώκουμε την εξουσία για την εξουσία, δεν θέλει κάτι τέτοιο ο Ουαταρά, αλλά θέλει να οικοδομήσει μια Κοντιβουάρ αρμονικά συνεργαζόμενη με τα κράτη σε μια δυτικοαφρικανική περιοχή που περιμένει τη συνεισφορά της στην περιφερειακή ολοκλήρωση μια χώρα η οποία να ενταχθεί αρμονικά στον κύκλο των δημοκρατικών χωρών. Βοηθήστε μας να μάθουμε τη δημοκρατία λοιπόν και να σεβαστούμε τους κανόνες της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Γραμματέα. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Τέλος της συνεδρίας σας.